Mes Καλημέρα και κύριοι. Είδατε όλη την ημερήσια διάταξη. Εφόσον δεν έχετε παρατηρήσεις θεωρείτε ότι είναι πλέον δεκτή. Έχω να κάνω διάφορες ανακοινώσεις από πλευράς της Προεδρίας. Σας έχουν διανεμηθεί διαθέσιμες γλώσσες. Γραπτός, δεν θα επανέλθω. Είναι κανονικές συνηθισμένε γλώσσες της Επιτροπής μας, γλώσσες εργασίας. Επίσης έχετε λάβει κάποια έγγραφα ή links για να βρείτε τα έγγραφα αυτά σε ηλεκτρονική μορφή, όπως σε όλες τις συνεδριάσεις μας. Επίσης πρέπει να πω ότι και αυτή η συνεδριασία είναι δημόσια και καλωσορίζω μια ομάδα επισκεπτών από τη ΜΚΟ Tax Justice Europe. Είναι 15 περίπου πρόσωπα επισκέπτες, τους οποίους έχω την ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίζω και να τους υποδεχόμαστε στις εργασίες μας και πραγματικά τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν αυτές τις δράσεις ενημέρωσης του Εβραίου κοινού για τις διάφορες ανομαλίες που διαπιστώνονται παγκοσμίω σε φορολογικά ζητήματα και κυρίως στην Ευρώπη. Η δράση η δική σας ε, βοηθάει και τη δικιά μας για να πείσουμε τις κυβερνήσεις να τερματίσουν ε, κάποιους ε, νόμους ή διοικητικές πρακτικές που για μας είναι απαράδεκτες. Και όπως όλες οι προηγούμενες δημόσιες συνεδριάσεις μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν έχουμε σημαντική συνεδρίαση που αφιερώνεται κυρίως στην ανταλλαγή απόψεων με τον Προεδρεύοντα ε, των κάτω χωρών που έχει την αρμοδιότητα ε, για τα φορολογικά. Ξέρετε ότι προεδρεύει στο πρώτο εξάμεινο η Ολλανδία και πριν έρθει ο υπουργό, θα ήθελα να σας κοινοποιήσω τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής μας των συντονιστών. Γνωρίζετε ότι υπάρχει σημαντικό πολιτικό ζήτημα που ετίθετο και έπρεπε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Το ποια θα ήταν δηλαδή τα πολιτικά αποτελέσματα και το πολιτικό προϊόν τρόπον τηνά της νέας αυτής επιτροπής τάξη 2. Δηλαδή, το, ετέθη το ερώτημα εάν θα καταλήξουμε σε έκθεση ή σε ψήφισμα. Ποια θα είναι η έκβαση και το τελικό προϊόν. Με συντριπτική πλειοψηφία οι συντονιστές θέλησαν ε, να συνταχθεί η έκθεση και να υποβληθεί στην Ολομέλεια κανονικά. Ένα οριστεί ε, όπως και την προηγούμενη φορά, όχι ένας αλλά δύο ε, συνεισηγητές, ο Κεπ Κόφωτ είναι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και ο Μίχαλ Τόιρερ από τους Ελευθέρους. Τώρα, ε, συγκρινόμενη η έκθεση με το ψήφισμα ενέχει μια υποχρέωση που σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Και η υποχρέωση είναι αυτή ότι σε όλα τα στάδια εργαζόμαστε σε όλες τις γλώσσες. Άρα χρειάζονται μεταφράσεις. Και όταν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, όταν το μετρήσαμε μάλλον αντίστροφα, διαπιστώσαμε ότι ήταν σχεδόν αδύνατο, ανέφικτο να γίνει έκθεση λόγω των διαφόρων ερευνητικών εργασιών που χρειάζεται για να συμπεριληφθούν τα στοιχεία στην έκθεση. Λέω λοιπόν ότι δεν προλαβαίναμε μέχρι την εκπνοή της ε, Επιτροπής μας που είναι η Δευτέρα Ιουνίου. Γιατί στις 2 Δεκεμβρίου αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων να ε, παρατείνει τις εργασίες, εν πάση περιπτώσει να συσταθεί μια δεύτερη Επιτροπή Τάξ με διάρκεια ζωής 6 μηνών. Γι' αυτό μου ανέθεσαν ε, οι εισηγητές να ζητήσω από τη διάσκεψη των Πρόεδρων μια τεχνική παράταση δίμηνη έτσι ώστε να μπορέσουμε σε περίπτωση που η διάσκεψη των Προέδρων το εγκρίνει έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα ε, το εγκρίνει για να καταθέσουμε ένα σχέδιο έκθεσης ενώπιον της Επιτροπής της 24 Μαΐου εδώ και να το ψηφίσουμε στη συνέχεια αφού συζητήσουμε τις τροπολογίες στις 20 Ιουνίου έτσι ώστε να πάει στην Ολομέλεια με το καλό τον Ιούλιο. Θέστηκα λοιπόν αντίστοιχη επιστολή στον πρόεδρο Σούλτ. Συμπληρώσαμε επίσης και επιβεβαιώσαμε τις προσκλήσεις που θέλαμε για τις ακροάσεις. για κοινέ εργασίες και για την αποστολή αντιπροσωπιών στο εξωτερικό. Για τις ακροάσεις. Ακούσαμε τον Επίτροπο Μοσκοβισή δύο φορές ήρθε σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ΕΚΟΝ. Σήμερα θα ακούσουμε την Ολλανδική Προεδρία για πρώτη φορά και σε περίπτωση που παραταθεί και η εντολή μας θα την ξανακούσουμε, θα σας πρότεινα, θα το δουν οι συντονιστές, αλλά αυτό θα τους προτείνω να ε, έρθει και στο τέλος της Προεδρίας της, η, Ολλανδική Προεδρία να μας ε, αναφέρει. Επίσης, έχουμε προβλέψει να ακούσουμε και άλλους δύο επιτρόπους που είναι η Επίτροπος Βεστάγκερ, αρμόδια για τον ανταγωνισμό που είχε έρθει και στην πρώτη για να ε, αρχίσουν να κινήσουν διαδικασίες για τις κρατικές φορολογικές ενισχύσεις που σύμφωνα με την άποψή της θεωρούνται λίγο σύμβατες με την ισότητα των ευκαιριών και τον ανταγωνισμό. 4 Απριλίου λοιπόν έχουμε προβλέψει να έρθει η κυρία Βέσταγκερ. Οι συντονιστές επίσης θέλησαν να ακούσουν τον Επίτροπο Λόρδο Χίλ που είναι αρμόδιες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα τραπεζικά. Και συμφωνεί και η Επιτροπή μας να δούμε σε μεγαλύτερο βάθος ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίζουν οι τράπεζες στις συμβουλές που παρέχουν στην πελατεία τους έτσι ώστε να διευκολύνουν κάποιες φορολογικές έτσι, κατασκευές την ακρόαση αυτή την κάνουμε και σε συνεργασία με εκπροσώπους των τραπεζών. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει για ημερομηνία για την ακρόαση ε, του Λόρδου Χίλ, διότι εκείνος είναι αρμόδιος για τις εκθέσεις αναχώρα και γύρω στα μέσα Απριλίου φαίνεται ότι θα καταθέσει το κείμενο αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος ε, Επίτροπος. Θέλει να έχει λοιπόν προηγουμένω την έγκριση τη εκτελεστική επιτροπή πριν έρθει ε, να μα παρουσιάσει το κείμενό του στη δική μα επιτροπή. Υπάρχουν και άλλε αρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, όπω η ΕΚΟΝ, η Γιούρη και θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τον τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει και η δική μας Επιτροπή να θέσει ερωτήσεις στο Λόρδο Χίλ μαζί με τους άλλους συναδέλφους σε αγαστή συνεργασία με αυτούς όπως συνήθως συμβαίνει. Για τις υπόλοιπες ακροάσεις προβλέπεται αυτή τη φορά αυτό το οποίο δεν είχαμε κάνει ή δεν είχαμε επαρκώς κάνει στην τάξη 1 θα υπάρξει ακρόαση των φορολογικών ειδικών δικαιοδοσιών ή κάπως ειδικών, πώς να το πω. Προβλέπεται για τις 14 Μαρτίου μια ακρόαση των τοπικών κυβερνήσεων του Γουένζε και του Τζέρσεϊ. Τους είχα συναντήσει εγώ σε προσωπικό επίπεδο εδώ και λίγους μήνες αλλά αυτή τη φορά θα έρθουν δημοσίως να μιλήσουν στο σύνολο της Επιτροπής Τάξ 2. Και τη 15η Μαρτίου ε, θα υπάρξει ακρόαση με τους εκπροσώπους της Ανδόρας, του Μονακό και του Λιχτενστάιν. Ε, θα είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται στις χώρες αυτές και σε ποιο βαθμό οι συστάσεις του ΟΣΑ στα πλαίσια του προγράμματος δράσης BEPS έχουν αλλάξει ή δεν έχουν αλλάξει το καθεστώς της συγκεκριμένης χώρας σε σχέση με τη φορολογία των επιχειρήσεων. Οι συντονιστές επίσης θέλησαν να προσκαλέσουν και αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις. αντιμετωπίσαμε την ίδια δυσκολία την οποία είχαμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει στα πλαίσια της τάξ 1. Επί τη βάση δηλαδή ποιων κριτηρίων θα προσκαλέσουμε κάποιες πολυεθνικές γνωρίζοντας ότι οι χρονικές διάρκειες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένες και γι' αυτό θα θέλαμε οι όποιες προσκλήσεις να οδηγήσουν σε ε, συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων με χρήσιμο τρόπο. Το κριτήριο των συντονιστών είναι να προσκληθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες στην παρούσα φάση υπόκεινται ε, διαδικασίες σε διαδικασίες ε, για φορολογικούς λόγους διαδικασίες οι οποίες έχουν προκληθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από τις διοικήσεις των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει επανάκληση επιχειρήσεων που έχουν ήδη έρθει εδώ και πιθανώς και κάποιες άλλες ήδη έχουν απευθυνθεί προσκλήσεις στην Google, την οποία έχουμε ήδη ακούσει και η οποία συμφώνησε, την Apple που συμφωνεί και αυτή την Fiat η οποία είχε αρνηθεί την προηγούμενη φορά και προς στιγμή δεν έχει απαντήσει. Την IKEA η οποία είχε έρθει την πρώτη φορά αλλά από τότε πήραμε νέες πληροφορίες και ευχαριστώ την ομάδα των Πρασίνων που είχε ζητήσει να διατυπωθεί, να συνταχθεί μάλλον μια πανεπιστημιακή μελέτη για την αρχιτεκτονική, τη φορολογική του Group IKEA και είχε πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε επίσης την απάντηση της επιχείρησης McDonald's που ήδη ακούσαμε την προηγούμενη φορά αλλά από τότε έχει ξεκινήσει εις βάρος της μία έρευνα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως επίσης και η ε, επιχείρηση Starbucks η οποία αρνήθηκε την πρόσκληση. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι ο τελικός. Αν υπάρξουν επιπλέον στοιχεία θα την συμπληρώσουμε σχετικά τώρα με το πιστοτικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η απόφαση η οποία έχει ληφθεί είναι σε συνεργασία με το Policy Department του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει μια κοινή secrétariat euh, d'un atelier σε συνεργασία λοιπόν με το Policy Department Α θα υπάρξει ένα, μια ομάδα εργασίας η οποία θα παρουσιάσει ερευνητικές ε, εκθέσεις ε, για το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα στα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, δηλαδή τα θέματα των ειδικών φορολογικών συμφωνιών ε, και θα ακολουθήσουν συναντήσεις με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων. Αντίθετα από τις ακροάσεις με πιστοτικά ιδρύματα που είχαμε κάνει στα πλαίσια του ΤΑΞ 1, είχαμε υποδεχθεί εκπροσώπους της BNP Paribas, της Barclays και της HBC, HCBC. Τώρα θα θέσουμε ερωτήσεις προς τις τράπεζες για τις σχέσεις τους με την πελατεία τους και για τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για μια καλύτερη ε, φορολογική στρατηγική τους πελάτες του. Έχουμε ακόμα έναν συγκεκριμένο αριθμό τραπεζών που θα θέλαμε να προσκαλέσουμε. Δεν το δημοσιοποιώ αυτό, διότι διαλόγου ευγενία θα ήθελα να προσκαλέσω πρώτα τους άμεσα ενδιαφερομένους πριν το ανακοινώσουμε δημόσια. Πρώτα δηλαδή θα πρέπει να πάρουν την πρόσκληση. Δεν θα πρέπει κάποιος υπεύθυνο μιας επιχείρησης να μάθει από τον τύπο ότι είναι προσκεκλημένος. Και όταν ολοκληρωθούν οι προσκλήσεις θα σας ενημερώσουμε. Αυτά για τις ακροάσεις. Προβλέπετε επίσης μια άλλη ακρόαση στα πλαίσια της συνάντησης των συντονιστών ε, διευρυμένη και με τα υπόλοιπα μέλη και με δημοσιογράφους και έχουμε την δυνατότητα να προσκαλέσουμε πολλούς από τους ε, δημοσιογράφους αυτούς σε μια δημόσια ακρόαση, σε μια τακτική μας συνεδρίαση. Ε, τώρα για τις αντιπροσωπείες, για τις επισκέψεις στο εξωτερικό προβλέπονται δύο αντιπροσωπείες. Η μία προβλέπεται για την Κύπρο είναι γνωστές οι ημερομηνίες 15 Απριλίου και έχουμε ένα σχέδιο προγράμματος το οποίο είναι ήδη στη διάθεσή σας. Και η άλλη αντιπροσωπεία έχει μεγάλη σημασία στη Washington την εβδομάδα της 16ης Μαΐου, αμέσως μετά δηλαδή την 50 ε, θα χρειαστούμε όλη την εργάσιμη εβδομάδα για να έρθουμε σε επαφή με τις Αμερικανικές Αρχές, με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Αμερικανικό Κογκρέσο και με την Επιτροπή Ways and Means, όπως επίσης και με την Finance Committee της Γερουσίας. Προσπαθούμε να κάνουμε μια συνεδρίαση από κοινού με τις δύο επιτροπές, θα κερδίσουμε χρόνο έτσι, έχει μεγάλη σημασία πόσο μάλλον οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο και το θέμα της φορολογίας είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητιώνται από τους υποψηφίους για την Προεδρία και το εν μέρει ανανεώσιμο Κογκρέσο. Και για την συνέχεια του προγράμματος δράσης BEPS έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρουν στις εσωτερικές τους νομοθετικές ρυθμίσεις τις συστάσεις του ΟΣΑ, αλλά και το ίδιο να κάνουν και οι υπόλοιποι εταίροι μας στον κόσμο, γιατί αλλιώς ε, τότε θα λειτουργήσουν οι συμφωνίες αυτές ε, εις βάρος μας και υπέρ αυτών. Εξάλλου και στα πλαίσια του ιδίου πνεύματος συνεργασίας με ένα μέγιστο αριθμό πολιτικών υπευθύνων σε σχέση με την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων τις οποίες έχουμε ήδη κάνει, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τρεις ε, διακοινοβουλευτικές συναντήσεις. Η μία από αυτές θα γίνει στις 18 Απριλίου με εκπροσώπους των 28 Εθνικών Κοινοβουλίων βάση εργασίας είναι το νομοθετικό πακέτο το οποίο έχει καταθέσει εδώ και λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο, Μοσκοβισή μας το παρουσίασε εδώ και λίγες μέρες και μετά μια συνάντηση στο Παρίσι σε συνεργασία και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΣΑ και την Επιτροπή Φορολογίας του ΟΣΑ θα είναι μια πρεμιέρα θα έλεγα γιατί θα υπάρξουν εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, 80 χώρες που συμμετέχουν στην προετοιμασία του προγράμματος δράσης BEPS για τον ΩΣΑ. Και τέλος, αυτό θα γίνει στις 2 Μαΐου. Και τέλος, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε, έχουμε το πρόγραμμα της Επιτροπής Ανάπτυξης Μαζί με την ΤΕΒΕ λοιπόν θα προσκαλέσουμε πάλι κοινοβουλευτικούς από τις υποανάπτυξη χώρες αυτή τη φορά για να ανταλλάξουμε μαζί τους πληροφορίες για τα προβλήματα και τις ζημίες που προκλήθηκαν στις χώρες αυτές από τις ε, ιδιαίτερα επιθετικές φορολογικές πρακτικές. Τέλος, Έχουμε περάσει στην τελική φάση, ήταν σχετικά περίπλοκο το θέμα μέχρι τώρα και για πολιτικούς λόγους αλλά και για διοικητικούς λόγους, αλλά είμαστε στην τελική φάση καθορισμού των προϋποθέσεων στα πλαίσια των οποίων η τεκμηρίωση την οποία ατελώς είχαμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα στα πλαίσια της tax 1, ιδιαίτερα σχετικά με τις εργασίες της ομάδας Code of Conduct, θα τεθούν τα στοιχεία αυτά στην διάθεση όλων των μελών της ΤΑΞ 2 με πολύ πιο ευρύ και αναλυτικό τρόπο και με πολύ πιο ευανάγνωστο τρόπο σε χώρους εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. θα πρέπει να αποφασίσουμε για κάποιες ε, πρακτικές λεπτομέρειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Τα έγγραφα όμως είναι ήδη στην διάθεσή μας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι συντονιστές έχουν ήδη ε, ε, έρθει σε επαφή και συζητήσει με τον νέο Γενικό Διευθυντή στο τέλος της συνάντησης ε, με το Γενικό Διευθυντή εμείς ε, ε, επαναλάβαμε τα, τον κατάλογο των εγγράφων για μια ακόμη φορά που έχουμε ανάγκη και θα πρέπει να μας επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες ότι εκτός από τα έγγραφα τα οποία ήδη είναι στη διάθεσή μας, ο κατάλογος τον οποίο έχουμε ζητήσει θα μας δοθεί εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί είναι προφανές ότι θα επιμείνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμβεί. Γνωρίζοντας βέβαια ότι ο Προεδρεύων Ολλανδός Υπουργός του ΕΚΟΦΗΝ, ο κύριος Βίμπες, ο οποίος θα έρθει όπου να είναι, είναι από πλευράς του υπεύθυνο για το θέμα αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου και γι' αυτό μπορεί να τεθεί το ερώτημα και προς αυτόν, ποια είναι η θέση του δηλαδή για το θέμα της πρόσβασης των κοινοβουλευτικών στα έγγραφα του Συμβουλίου γενικότερα και στα πρακτικά των συνεδριών της Γραμματείας του Συμβουλίου σε επίπεδο COC. Νομίζω ότι το Συμβούλιο ε, θα επιδείξει μεγαλύτερη δεκτικότητα από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Ε, αυτά έχω αγαπητοί συνάδελφοι να σας πω. Ε, μακρηγόρησα λίγο αλλά έχει ζητήσει το λόγο Σβέν. Ε, σας ευχαριστώ για μια πλήρη παρουσίαση και ιδιαίτερα αναλυτική των στοιχείων θα ήθελα να πω ότι από την ίδια συνάντηση των συντονιστών θα ήθελα να μοιραστώ κάτι με τους συναδέλφους. Όπως έχει ήδη υποθεί υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Διεύθυνση ΚΟΜΠ. Συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο γιατί πρέπει να χαιρετήσω, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, μάθαμε στα πλαίσια της συνάντησης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις δυνατότητες να παρακολουθήσει κάποιες περιπτώσεις φορολογικών παρεμβάσεων κρατικών. Μετά λοιπόν και επί τη βάση των αποφάσεων των δικαστικών για ορισμένες γνωστές αποφάσεις, για να παρακολουθηθούν από κοντά και να εξεταστούν τα θέματα αυτά και να ζητηθεί επιστροφή της ε, μη δέουσας αληθής ε, ε, επιδότησης είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παράφορη, κατάφορη μάλλον, παραβίαση των νομιθετικών ρυθμίσεων. Γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να συνεχίσουν να παίρνουν τα πλεονεκτήματα τα φορολογικά τα οποία είχαν στο παρελθόν και νομίζω ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι και για την ισότητα μπροστά στον νόμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού να μην διασφαλίσει την ισότητα μπροστά στον νόμο και να μην διεκδικήσει την επιστροφή όλων των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έχουν δοθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ συνάδελφε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Το αναφέρατε και σε επίπεδο συντονιστών και είμαι βέβαιος ότι οι συγητές θα αναφερθούν σε αυτά όλα. Χαιρετώ λοιπόν και ευχαριστώ για την παρουσία του τον Υπουργό Βίμπες ο οποίος είναι ο υπεύθυνος υπουργός για θέματα οικονομικών και φορολογικών στην Ολλανδική κυβέρνηση. Με χαρά σας συναντάμε εκ νέου. Σας είχαμε συναντήσει εδώ και λίγους μήνες κύριε Υπουργέ. Στη Χάγη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης την οποία έκανε η Επιτροπή μας στην χώρα σας, όπως επίσης και σε άλλες 5-6 ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε ιδιαιτέρως ε, ε, ενδιαφέρον θα ακούσουμε από πλευρά σας το πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου το οποίο θα είναι καθοριστικό για τα θέματα τα οποία συζητάμε. Ιδιαίτερα μετά από το πακέτο το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε σαν συνέχεια των συστάσεων του προγράμματος δράσης BEPS του ΩΣΑ. Και ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η θέση της Ολλανδικής Προεδρίας για το CCCTB, όπως επίσης και για τα μέτρα γυτνίασης και συνδυασμού των φορολογικών μέτρων για τις επιχειρήσεις. Αυτά όλα βρίσκονται σε επίπεδο προπαρασκευαστικό στην Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι και είδατε ότι σε αυτούς τους δύο τομείς η Επιτροπή Τάξ 1 κατέθεσε μια σειρά συστάσεων και εκτιμούμε ιδιαίτερο τις απόψεις της Ολλανδικής Προεδρίας επί των συστάσεων αυτών. Παρ' όλα αυτά θα σας τεθούν και ερωτήσεις για την παρακολούθηση ή μάλλον για τη συνέχεια την οποία η Ολλανδική Προεδρία, που είναι υπεύθυνη για την Προεδρία του Συμβουλίου στην παρούσα φάση, έχει δώσει ή θα ξεκινήσει να δίδει στις συστάσεις αυτές. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν για να κάνετε μια δεκάλυπτη περίπου εισαγωγή και στη συνέχεια οι συνάδελφοι θα σας θέσουν ερωτήσεις σε πεντάλεπτο ερώτηση και απάντηση μαζί. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο parole. Does this work? Yeah. Δουλεύει το μικρόφωνο, ναι. Καταρχά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση ω Προεδρία του Συμβουλίου σε αυτή την άτυπη ανταλλαγή απόψεων για κάποια θέματα φορολογικού χαρακτήρα. Θα δεχτείτε ε, τη συνήθεια που έχω από το Eurogroup που να μιλώ αγγλικά. Ε, όπως έχει τονιστεί και στη δική σας έκθεση, η αντιμετώπιση ανεπιθύμητης ε, και επιθετικής ε, φορολογικής δράσης από πλευράς πολυεθνικών ήταν πολύ ψηλά στο θεματολόγιο και στις προτεραιότητες και του ΟΣΑ και της ομάδας των 20. Θα συνεχίσει η Προεδρία των Κάτω Χωρών την εργασία που άρχισε επί Λουξεμβουριανής Προεδρίας που έχει κάνει παντιέρα της στο θέμα το, ε, αυτό της καταπολέμησης φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη του ε, Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών ΕΚΟΦΗΝ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου είδαμε ότι έχει γίνει δουλειά και έχει ολοκληρωθεί στον ΟΣΑ και στο G20 και το Συμβούλιο έχει διατρανώσει την επιθυμία του να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και στην συνέχιση που θα δοθεί ιδιαίτερα στις αποφάσεις για το ΠΕΠΣ που είναι η διάβρωση της βάσης και η μετατόπιση των κερδών. Η προτεραιότητα θα γίνει ε, με πραγματική νομοθετική προσπάθεια ε, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε αυτή την έκκληση καταθέτοντας ε, τον Ιανουάριο ε, την δέσμη μέτρων για την ε, αποφυγή φορολόγησης, ΑΤΑΠ είναι τα αρχικά, για να διαρθρωθεί και να δομηθεί κάπως η δουλειά στο Συμβούλιο. Έχουμε προετοιμάσει αντίστοιχο έγγραφο και οδικό χάρτη, είμαι βέβαιος ότι το έχετε δει, με συγκεκριμένες δράσεις για να κατα πολεμηθεί το BEPS, που είναι η διάβρωση της βάσης και η μετατόπιση των κερδών. Και τα μέτρα αυτά θα προωθηθούν στο Συμβούλιο βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και μάκρο πρόθεσμα. Συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν θα γίνουν για τα διάφορα θέματα που είναι επιτάπητο στο Συμβούλιο. Specifically, we'll seek rapid progress on some of the ε, στα θέματα BEPS θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, όπως ε, είναι η οδηγία για την αποφυγή της φορολογίας, αλλά και την οδηγία ε, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, το DAC 4 που ονομάζεται, και θέλουμε να αναθεωρήσουμε και τον κώδικα δεοντολογίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Οι συζητήσεις του πρόσφατο ECOFIN έδειξαν πόσο δύσκολη είναι η φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο προβληματική, αλλά είναι και πρόκληση. Είδαμε ένα ακρό φάσμα από τη μια μέχρι την άλλη πλευρά ή την άλλη άκρη. Και υπάρχουν και χώρες που έχουν ειδικέ θέσεις και ειδικά προνόμια και κίνητρα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα έσοδα από τη φορολογία αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέρη της Ευρώπης παραμένουν ε, ελκυστικά για τις επενδύσεις. Θα γνωρίζετε ότι σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για μεμονωμένα κράτη-μέλη και καθεστώτα φορολογικά που ισχύουν εκεί ούτε καν για το ίδιο το Ολλανδικό. Αλλά με χαρά να ανταλλάξουμε απόψεις για το τι ε, κάνουμε στο Συμβούλιο και τι πρόκειται και προτιθέμεθα να πράξουμε μέχρι τα τέλη της ε, Προεδρία των Κατοχωρών. Καταρχά. να δούμε μερικέ από τις προτεραιότητε. Για παράδειγμα, η έκθεση αναχώρα και το DAC 4, η σχετική οδηγία. Η Ολλανδική Προεδρία έχει την πρόθεση να ε, καταλήξει σε μια ε, πολιτική ε, συμφωνία και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες αυτό το καιρό. Υπάρχουν μεταξύ ημών άνθρωποι εδώ παρόντες που έχουν αφαιρώσει πάρα πολύ χρόνο, μέρες ολόκληρες για τη συμφωνία. Έχουμε την πρόθεση να φτάσει αυτό το θέμα στο εκοφήν του Μαρτίου, ε, έχοντας ήδη την προοπτική μιας πολιτικής συμφωνίας από το Μάρτιο. Ελπίζω αυτό να στεφτεί με επιτυχία. Και τώρα ε, θέλουμε να έχουμε και τη γνωμοδότηση και προσβλέπουμε στη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλο θέμα είναι η οδηγία για ε, την ε, καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Αντίστοιχη προσέγγιση και θέλουμε να υπάρξει μια σύντομη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Έχουν αρχίσει οι διεργασίες για να συμφωνήσουμε το συντομότερο δυνατό. Και στην ε, προεδρία αυτή βεβαίως πριν ολοκληρωθεί, πριν το καλοκαίρι. Ε, άλλο θέμα είναι η οδηγία ε, για για τα δικαιώματα χρήσης και τα επιτόκια. Για την ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας επίση, πρέπει να σας πω ότι συνεχίζει να μα απασχολεί το ε, μέλλον του κώδικα, δηλαδή πώς θα γίνεται η διακυβέρνηση, η διαχείρισή του και προτείνονται μέτρα για την ενίσχυση στο μέλλον, λαμβάνοντα υπόψη την επιθυμία του ΕΚΟΦΗΝ στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου να βρεθεί ε, μια παραδεκτή ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση της ε, διαφάνειας της ομάδας εργασίας από τη μια και τη διατήρηση ε, της ε, απόρριτης ε, φύσης των εργασιών. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση, βεβαίως με μύθια να συζητούμε κάποια θέματα, αλλά ταυτόχρονα να ενημερώνουμε με δημοκρατικό τρόπο για το τι συμβαίνει. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης μέγιστη διαφάνεια, αλίμονο, έτσι ώστε να, οι συζητήσεις να γίνονται προσανατολισμένες πάντα σε αποτελέσματα. Ως Προεδρία επίσης ε, ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις απάτες ε, που συνδέονται με το ΦΠΑ. Μπορεί να μην είναι το αμέσου ενδιαφέρον αλλά ο όγκος είναι πολύ μεγαλύτερος στο φόρο προς τις αξίες από ό,τι στα κέρδη. Και υπάρχουν παντού ευκαιρίες για απάτη και αξίζει τον κόπο να μελετηθεί. Είναι προτεραιότητα για την Προεδρία των Κάτω Χωρών και πέρα από τα παραδοσιακά υφιστάμενα μέτρα θα πρέπει να κοιτάξουμε να θεσπίσουμε πιο καινοτόμα. Και από τα αγαπημένα μου είναι η χρήση ανάλυσης, ε, ε, μάλλον δικτύου ανάλυσης συναλλαγών. Αυτό ε, το, έχουμε ήδη αναπτύξει στην Ολλανδία και μπορούμε να συνδυάσουμε όλη τη γνώση υφισταμένων δικτύων που παρακολουθούν την απάτη με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΦΠΑ με τρόπο ευφύ μπορεί να γίνει αυτό χωρίς ε, ε, ιδιαίτερα αγκητικό φόρτο μεγάλο για τις καλόπιστες επιχειρήσεις. Και μπορεί κανείς να εντοπίσει την απάτη, την ενδεχόμενη πριν καν συμβεί. Ε, θα, θα πω αυτά στο ΕΚΟΦΗΝ και θα προσπαθήσω να πείσω τα μέλη του Συμβουλίου ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με αυτό. Επίσης, ε, θέλουμε να δούμε και άλλα μέτρα καταπολέμησης ε, Τη απάτη και ενδεχομένω και πιλωτικά προγράμματα για να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απάτη αυτή στο φόρο της αξία πάντα. Τώρα, η Ολλανδική Προεδρία έχει πλήρη επίγνωση τη ανάγκη ότι πρέπει να επιτευχθεί πρόοδο στη φοροαπηφυγή και στη φοροδιαφυγή στην καταπολέμησή του. Δηλαδή, θα πρέπει να προχωρήσουμε και έχουμε ήδη προχωρήσει με πάρα πολλοί ταχυδισμού πιο γοργού από ποτέ. Επαναλαμβάνω, είμαστε προσιλωμένοι στην ε, κατεύθυνση αυτή. Στο κοφή θα το φέρουμε το θέμα της φορολογίας ε, με τρόπο αποτελεσματικό, πλήρη και ε, προσπαθώντας πάντα να επιτυχάνουμε συνένεση για κάποια θέματα. Και υπό την έννοια αυτή και υπό το πνεύμα όλων αυτών με ενδιαφέρον θα ακούσω τις απόψεις σήμερα. Ευχαριστούμε Υπουργέ αναφερθήκατε στον ΦΠΑ. Δεν έχουμε ευθυσουσίας αρμοδιότητα για το θέμα αυτό στην τάξη 2. Αντιθέτως, η ΕΚΟΝ αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση για αυτό το ζήτημα και σίγουρα θα εισακουστείτε με ιδιαίτερη προσοχή. Θα περάσω τώρα στον κατάλογο των ομιλητών και όπως σας είπα όπως και στις περισσότερες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ήθιστε ανάμεσα ε, για κάθε ε, συνδιαλλαγή ανάμεσα στον προσκεκλημένο και στο μέλο της Επιτροπή δεν υπερβαίνει το πεντάλεπτο. Παρακαλώ να μην υπερβαίνετε λοιπόν το χρόνο αγόρευση, ούτω ώστε να έχει στο, στη διάθεσή του Υπουργό ο χρόνο να μα απαντήσει. Αρχίζουμε από του δύο συνεισηγητέ. Γέπε Κόφοντ από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Βίψ, εδώ είμαι αριστερά. Θα ήθελα να πω ότι μας ευχαριστεί ιδιαίτερος που ήρθατε για τη σημερινή συζήτηση. Οι σοσιαλιστές ε, ε, και οι δημοκράτες ενδιαφέρονται όλους ιδιαίτερως για το πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας, κυρίως για το θέμα της ε, αποτελεσματικής εφορολόγησης, της φορολογικής διαφάνειας και του φόρου επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα ήθελα να επεκταθείτε για το χρονοδιάγραμμα. Αναφερθήκατε σε κάποιες φιλοδοξίες της Ολλανδικής Προεδρίας, θα ήθελα όμως να επεκταθείτε ή δυνατόν για το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να γίνω τα εξή ζητήματα. Η έκθεση αναχώρα ε, το CCR, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα ε, που ε, μας απασχολεί εδώ καιρό και είπατε ότι θέλετε να περιμένετε την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν όντω κάνει θετική αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και είναι αναμενόμενο, θέλουμε να ξέρουμε θα προωθήσετε το ζήτημα, ούτω ώστε να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των εκθέσεων ανά χώρα. Νομίζω ότι για το Κοινοβούλιο και γενικότερα για την Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το ζήτημα. Θα το προωθήσετε το ζήτημα και με ποιο τρόπο. Κατόπιν, Αναφερθήκατε στην ομάδα κώδικα διοντολογίας. Χαίρομαι που αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα και είπατε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ως προς τη διαφάνεια και ως προς την εντολή θα έλεγα εγώ θα προσέθετα ούτως ώστε να μπορέσει να επιληθεί άλλων ζητημάτων η ομάδα. Ε, κυκλοφορούν φήμες, γίνονται συζητήσεις ότι το Συμβούλιο έχει ήδη ε, συζητήσει διεξοδικά αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αν έχουν αναλυφθεί αποφάσεις, αν έχουν δρομολογηθεί αποφάσεις σε σχέση με αυτήν την ομάδα κώδικα διοντολογία ούτω ώστε να είναι, γίνει αποτελεσματική και να καταστεί διαφανέστερη αυτή η Επιτροπή. Αν δούμε ιστορικά τι έχει συμβεί στις κάτω χώρες, Και βλέποντας και τι συμβαίνει τώρα, αν δούμε το 2005-2007 παραδείγματος χάρη, κάποια περιστατικά. Ξέρουμε ότι η χώρα σας έχει αντισταθεί σε κάποια σημαντικά βήματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ποια είναι η στάση σας για αυτό το ζήτημα, ο υπουργό. Λοιπόν, έκθεση αναχώρα και η δημοσιοποίηση των εκθέσεων. Αυτή ήταν η πρώτη σας ερώτηση. Ναι τηρούσε η κυβέρνησή μου τη στάση ε, πως ε, δεν θα έπρεπε να αποφασίσουμε πριν από την πλήρη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μια ισχυρή επιθυμία για, την, για τις δημόσιες εκθέσεις ο ρόλος της Προεδρίας είναι να προωθεί το ζήτημα για να επιτευχθεί συντονισμός και όχι να τάσεται σε, στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Εάν λοιπόν είναι θετική εξελόγηση θα ταχθούμε υπέρ, αλλά όταν κάποιος ε, έχει την Προεδρία το ζητούμενο δεν είναι να τοποθετηθεί, το ζητούμενο είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και αυτό θα κάνουμε και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεδομένου το χρονοδιαγράμματος, γιατί στην αρχή νομίζω ήταν ένα και καλυμμένο επιπρόσθετο ερώτημά σας, έχω την... Ε, ε, ο στόχος μας, ναι, όντως είναι να καταλήξουμε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αλλά ε, πρώτα πρέπει να δούμε την αξιολόγηση και να ξεκινήσει ο διάλογος. Είπατε ότι δεν είναι απίθανο να είναι θετική η αξιολόγηση. Θα συμφωνήσω με τις προσδοκίες αυτές. Για την ομάδα COC, κώδικα διοντολογίας, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Πρώτον, η εντολή. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο προς το παρόν αν τροποποίηση της εντολής ε, θα οδηγήσει ε, σε νέα μορφή αυτής της ομάδας, σε νέα εντολή και σε περισσότερη διαφάνεια, θα δούμε. Και επειδή ένα ε, πιο δημοφιλές ζήτημα είναι αυτό της διαφάνειας, θα ήθελα να προσθέσω ότι Θα ήταν καλό να υπάρχει πιο εμπεριστατωμένη υποβολή ε, των στοιχείων μετά από τις ε, διαβουλεύσεις αυτής της Επιτροπής, μιλώντας και για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα επιδιώκουμε φυσικά, όμως προς το παρόν δεν έχουν στεφθεί με επιτυχία αυτές οι προσπάθειες. Δεν υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου και δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε. Ε, πάντως, ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα πιέσουμε. Θέλουμε να σημειωθεί η πρόοδος. Ευχαριστώ, κύριος Λαμασούρ. Για αυτό το τελευταίο που είπατε, Υπουργέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για την Επιτροπή Τάξης και μας εξέπληξε το ότι μέχρι στιγμή τα έγγραφα εργασίας της ομάδας COC που μας διαβιβάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ήταν διαβαθμισμένα ήταν λογοκριμένα και αυτό οφειλόταν στο ότι οι μισές χώρες δεν ήθελαν να δημοσιοποιηθούν ε, τα έγγραφα, να δοθεί πρόσβαση στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή και η Ολλανδία ήταν από τις χώρες που δεν επιτρέπανε την αποκάλυψη αυτών των ε, εγγράφων εργασίας και νομίζω ότι είναι λυπηρό διότι σώμαστε όλοι ε, υπέρ της διαφάνειας και σίγουρα θα ακούσετε αυτά τα ερωτήματα περί διαφάνειας και από άλλους συναδέλφους. Ο Μιχαήλ Τόιρερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος της Ομαδικής Προεδρίας, σας ευχαριστώ καταρχάς ε, που ήρθατε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να επιτευχθούν ε, πρόοδοι σε αυτό το τομέα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Γνωρίζετε ότι στην έκθεση τάξη 1 που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο απευθύνθησαν κάποιες συστάσεις και θέλω να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Ε, στο BEPS ακούμε ότι θέλετε να κάνετε δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό είναι βασικό στοιχείο ε, της έκθεσής μας ότι ο συνδυασμός 28 περίπλοκων φορολογικών συστημάτων δημιουργεί παραθυράκια που μπορούν να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν ε, για να πληρώσουν λιγότερους ή καθόλου φόρους κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ε, και σε σχέση με αυτό αποκομίσαμε την εντύπωση ότι η Ολλανδική Προεδρία εδώ έχει την πρόθεση να δράσει. Υπάρχουν όμως τώρα κάποια μηνύματα ε, σε ό,τι αφορά ε, τη δεσμευτική ε, νομοθεσία ότι η καινοτομία και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ευρεσιτεχνίες δεν θα είναι ε, στοιχείο αυτού το patent, patent boxes. Πώς το βλέπετε και μπορείτε να μας το διευκρινίσετε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Δεύτερον, πώς θέλετε να αποφύγετε μελλοντικά να μετατοπιστούν τα κέρδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, χώρες με χαμηλή φορολογία και μηδενική, στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. Μόλις πριν από λίγες μέρες είδαμε δημοσιεύματα για μια έκθεση που αν κατάλαβα καλά η Google περίπου σύμφωνα με δικά τη στοιχεία έχει μεταφέρει 11 δισεκατομμύρια ευρώ στις Βερμούδες υποτίθεται με ένα νόμιμο κατασκεύασμα και τα έχει μεταφέρει στις Βερμούδες. Ε, αυτά πώς θα βλέπει η Ολλανδική Προεδρία έτσι ώστε στο μέλλον να αποφεύγονται τέτοια φορολογικά κατασκευάσματα και μοντέλα. Ευχαριστώ. Πηγαίνω στην Ολλανδία. Πηγαίνω στην Ολλανδία αντί να πηγαίνω. Um, let me first... Θα ήθελα να ανταποκριθώ ε, πρώτα σε ανησυχίες ε, του Προέδρου. Είπατε ότι κάποιες χώρες δεν αποκάλυψαν ε, κάποιες πληροφορίες στο παρελθόν. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς την Επιτροπή Κώδικα Διοντολογίας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες ρυθμίσεις για την εμπιστευτικότητα και πρέπει να τηρηθούν. Ταυτόχρονα όμως υποχρεούμαστε να λειτουργούμε διαφανέστερα για το μέλλον και είναι με δέσμευση της Ολλανδίας προς αυτή την κατεύθυνση διότι ναι και τώρα θα αλλάξω καπέλα και θα μιλήσω εξ ονόματος της Ολλανδίας η χώρα μας θέλει να τηρεί τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, εγώ έχουμε κλείσει, όχι μόνο σε επίπεδο κειμένης αλλά και στη Βουλή μας. είναι ε, ξεκάθαρη ταυτόχρονα η επιθυμία να επικρατήσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει, ήθελα να το διευκρινίσω λοιπόν. Κύριε Τόερερ. Είπατε ότι ακούσατε κάποιες εφήμες ότι δεν συζητούνται καν τα patent boxes ε, για τα ευνοϊκότερα καθεστώτα, δηλαδή για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τι εννοείτε. Ε, διακόπτω κύριο Στόιρερ. Ε, ακούσαμε ότι δεν θα υπάρξει δεσμευτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνής και για την κοινοτομία. Αληθεύει. Δεν ξέρω που τα ακούσατε, απαντά ο υπουργό, που πάντως Με αυτά τα patent boxes, ε, τι συμβαίνει, πολλές χώρες ε, αναγκάζονται να τροποποιήσουν ε, τα δικά τους καθεστώτα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για να ευθυγραμμιστούν με την πρακτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέτος έχουν αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Πολλά συμβαίνουν λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις για τα διπλώματα ευρεσέχνες. Πολλές χώρες πρέπει να τροποποιήσουν τα καθεστώτα τους. Ξέρω γιατί, από πού πηγάζει αυτή η ανησυχία, διότι ε, ακούω τέτοιες φήμες, όμως σημειώνεται με μεγάλη πρόοδος. Ε, μεταβίβαση κερδών προς φορολογικούς παραδείσους μετά. Είναι ξεκάθαρο πως αν ε, υπάρχει μια φοροαποφυγή θα χρειαστεί να ληφθούν, να μέτρα κατά της ε, φοροαποφυγής. Υπάρχουν τέτοια μέτρα στο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πρόσφατο παρελθόν εγκρίναμε μια σειρά από μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μετατοπίζονται τα κέρδη ε, για φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Ο κύριος Τόιρερ, ένα λεπτό, μία επερώτηση. Κατάλαβα καλά, ε, πρόεδρε, ότι υποστηρίζεται την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την θέσπιση νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα patent boxes ε, ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνής και για την καινοτομία. Κατάλαβα καλά την απάντησή σας. Απάντηση. Πέρυσι και στην Επιτροπή ΚΟΚ και στον ΩΣΑ βρήκαμε ένα τρόπο για να μεταρρυθμίσουμε τα διπλώματα ευρεστέχνειας, τα καθεστώτα δηλαδή για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Μιλάτε για συγκεκριμένες οδηγίες, ναι, έχει ρυθμιστεί, έχει διεκπαιρεωθεί το ζήτημα. Το έχουμε ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε όντω, αλλά έχει ρυθμιστεί. Ο κύριος Λαμασούρ απαντάει, άρα είναι καταφατική η απάντηση ή υπάρχει παρανόηση. Τέλο πάντων θα εξετάσουμε εξωδικότερα το ζήτημα. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που είχαμε προβλέψει για τους συνεισηγητές. Παρακαλώ να μην υπερβαίνετε τα πεντάλεπτα εφ' εξής. Ε, Ελκ Χιμπνερ Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα και ευχαριστώ, αν κατάλαβα καλά, που είπατε πως η Ολλανδική Προεδρία δεν πιέζει μόνο για την εκπόνηση νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχετε και βαθιά κατανόηση σε σχέση με την πρώτη που πρέπει να σημειωθεί και σε επίπεδο soft law. Ε, υπάρχουν δύο έγγραφα στο τελευταίο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέσα στην ανακοίνωση. Ε, ένα είναι ε, πολιτική την εξωτερική πολιτική για τη φορολόγηση, κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται αξιολόγηση από πλευρά τη Επιτροπή σε σχέση με το αν συμμορφούνται ναι ή όχι με του κανόνε καλή ε, διακυβέρνηση ε, μία χώρα. Βεβαίω δεν υπάρχουν μέτρα κυρώσει που να προβλέπονται ε, κατά αυτών των χωρών και δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια ε, περαιτέρω προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερον, όταν μιλάμε για το καθεστώς μόνιμης εγκατάστασης, ε, δηλαδή ε, τεχνητή αποφυγή του καθεστώτους ε, ε, μόνιμης εγκατάστασης. Ξέρετε ότι στο BEPS προβλέπει όσα τροποποίηση του άρθρου 7 της σύγχρονης ευρωλογικής σύμβασης για να αποφευθεί η τεχνητή αποφυγή του καθεστώτος μόνιμης εγκατάστασης. Υπάρχουν σε αυτό το άρθρο 5 στο τροποποιημένο άρθρο 5 της Έμβασης σε συγκεκριμένα μέτρα. την ανακοίνωση του Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν ε, τη νέα διάταξη του εν λόγω άρθρου 5 στις ε, φορολογικές συμβάσεις ε, που διαπραγματεύονται διμερώς με συγκεκριμένα κράτη, τρίτες χώρες και ευελπιστεί έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτή την τεχνητή αποφυγή μόνιμη εγκατάσταση. Στη συνέχεια τέλη Νοεμβρίου είχαμε όμως ε, και το, τη στάση το έγγραφο της Λουξεμβουριανής Προεδρίας, το ενοποιημένο κείμενο και ήταν κατά τι διαφορετική η προσέγγιση για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ε, πρότεινε η Λουξεμβουριανή Προεδρία να συμπεριληφθεί στην οδηγία για ένα άρθρο, δηλαδή να μην περάσουμε μέσα από τροποποίηση των διμερών συμφωνιών των κρατών μελών με τρίτες χώρες, αλλά να σχετιστεί αυτό με την οδηγία για το BEPS. Τι θα κάνει λοιπόν η Επιτροπή, ε, ε, το Συμβούλιο, συγγνώμη, Ολλανδική Προεδρία, θα ακολουθήσετε τη γραμμή του ενοποιημένου εγγράφου της Λουξεμβουργιανής ε, Προεδρίας σε σχέση με το split της CCTB ή θα ακολουθήσετε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απάντηση για το θέμα της μόνιμης εγκατάστασης και της αποφυγής του καθεστώτος, από όσο καταλαβαίνω, ο ΣΑ εξέδωσε μία σύσταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μετέτραψε επίσης σε σύσταση. Άρα είναι μέρος του πακέτου και των διαπραγματεύσεων. Εάν σε με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις, θα έχουμε και συμπεράσματα του Συμβουλίου. Όμως δεν μπορούμε να τα εφήβρουμε αν δεν υπάρχουν ακόμη, είναι μέρος του πακέτου και επεξεργαζόμαστε αυτή τη σύσταση. Επίσης, κυρία Χίπνερ, λυπάμαι, αλλά δεν κατανοείς ακριβώς την πρώτη σας ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χιούμπνερ, ε, ρώτησα αν έχετε συγκεκριμένη στάση σε σχέση με τη χρήση των, ε, του soft law ε, Δηλαδή, ανακοίνωση παραδείγματο χάρη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, του Ιανουαρίου για την ε, εξωτερική πολιτική φορολόγηση. αυτή την ανακοίνωση υπάρχουν κριτήρια που προσδιορίζονται και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται η αξιολόγηση σε σχέση με το αν ε, τηρεί τα πρότυπα χρήστη διακυβέρνηση σε ένα κράτο. Όταν μιλάμε για τι non-cooperative jurisdiction, δικαιοδοτικέ αρχέ που δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Αυτά τα κριτήρια, εάν δεν πληρούνται, τι θα κάνει το Συμβούλιο, θα το διαπιστώσει και θα προχωρήσει χωρίς να επιβάλλει κάποια μέτρα. Αυτό ρώτησα. commission... Η Επιτροπή εκπονεί πρότασης για να συμπεριληφθούν τέτοιες ρήτρε σε άλλες συμφωνίες ε, με τρίτε χώρες και επίσης ε, εκπονεί και κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση των χωρών ε, για φορολογικούς σκοπούς ούτως ώστε ο δεσμός ανάμεσα στην αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επίπεδο καλή διακυβέρνηση αυτών των κρατών μελών να συνδεθούν. Είναι αρκετά δραστικό αυτό το μέτρο. Λοιπόν, προβλέπετε ότι κάποια στιγμή θα προκύψουν συμπεράσματα του Συμβουλίου και ενδεχομένως να επιληφθεί του ζητήματος και η Επιτροπή Κώδικα Διοντολογίας, COC. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ουγ Μπαγιέ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Euh, euh, Ευχαριστώ που είστε εδώ κύριε Υπουργέ. Να επανέλθω στην προηγούμενη οδηγία για τη διαφύγη. <clears throat> Στο Συμβούλιο κάποιες χωρεμέλη θα ήθελαν να περιοριστούν σε ένα κείμενο το οποίο να προέρχεται άμεσα και ε, χωρίς περισσότερα στοιχεία από το BEPS. Ε Ενώ ο ίδιος ο κύριος Μοσκοβισή είχε αδιαφερθεί και στο λεγόμενο switch over, όπως επίσης και στον γενικότερο κανόνα για τις καταχρήσεις, κατά των καταχρήσεων. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα επιμέρους στοιχεία στο κείμενο, τότε το κείμενο αυτό δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάσταση. Τι ακριβώς γίνεται, υπάρχει μια διαίρεση μεταξύ σας ή μπορείτε να τα συζητήσετε σε επίπεδο κρατών μελών. Δεύτερη ερώτηση. Άκουσα ότι έχετε προχωρήσει <clears throat> για το patent box, τα ευνοϊκά καθεστώτα για διπλώματα ευαισθηχνίας, αλλά στο βασικό κείμενο δεν υπάρχει ορισμός. Εάν θέλουμε πράγματι να καταπολεμήσουμε κάτι, πρέπει να συμφωνούμε σε ένα κοινό ορισμό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μέχρι τώρα μπορείτε να καταλήξετε σε μια κοινή προσπάθεια ορισμού. Και τώρα ένα θέμα το οποίο έχει σχέση περισσότερο με τη δική σας χώρα. Δεν θα έρθω στα θέματα των δεσμών και του CCTB. Ξέρουμε τι έγινε μετά από τα Swiss Leaks και τα Lux Leaks. Ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η χώρα σας είναι από αυτές που δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα πρόθυμη, μαζί με άλλες βέβαια. Φοβάμαι ότι ώσπου να συμφωνήσουν όλοι δεν θα υπάρξουν εκείνα βήματα. Ε, τι παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε η δική σας χώρα να μην έχει μέχρι τώρα αποφασίσει να πάρει μέρος. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Μπαγιέ, Έχω ένα πρόβλημα με τις ερωτήσεις σας, γιατί εσείς αναφερθήκατε και στο CCTB και στην ρήτρα switchover ε, και στα FTT και στα patent boxes. <clears throat> Κάποια από τα θέματα αυτά είναι σαφώς υποσυζήτηση και εγώ είπα ήδη ότι η Ολλανδική Προεδρία θέλει να οδηγηθούμε σε μια κάποια συμφωνία. Είμαστε κοντά για την Retra Switchover είναι τμήμα του λεγόμενου πακέτου ATAP. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί επί μακρόν στις διάφορες ομάδες εργασίας και στο ΕΚΟΦΗΝ. Το CCCTB, η κοινή βάση, δεν είναι υποσυζήτηση στην παρούσα φάση. Δεν υπάρχει ε, επί του παρόντος πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την Ολλανδική Προεδρία θα έχουμε προτάσεις, οπότε δεν είναι δυνατόν να γνωμοδοτήσω εγώ. Βέβαια σαν εκπρόσωπος της χώρας μου μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου, αλλά δεν είμαι γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μου δημιούργησαν οι ερωτήσεις σας κάποια σύγχυση. Πάντως το ATAP και το switch over έχουμε προχωρήσει και θα είναι μέσα στη συμφωνία και ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Δουλεύουμε γι' αυτό με σκληρό τρόπο. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι Ολλανδοί δεν είναι τμήμα των χωρών που συζητούν το FTT, τον φόρο αυτό επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτό όμως δεν εμποδίζει και κανέναν άλλον να κάνει κάτι αν θέλει να το προχωρήσει. Κανένας δεν θα περιμένει είτε την Προεδρία είτε τους Ολλανδούς. Δεν βλέπω πού υπάρχει πρόβλημα. The question was why. Το ερώτημα είναι γιατί αν έχω ακόμα 30 δεύτερα. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Εργάζεστε για να καταλήξετε σε ένα κοινό ορισμό της μόνιμης εγκατάστασης και των ε, τιμών ε, μεταβίβασης. Γιατί δεν υπάρχει κοινό ορισμό. Τι συζητάτε. Ε, δεύτερο. Και τελευταία ερώτηση δεν απαντήσατε. Για ποιο λόγο οι κάτω χώρε δεν θέλουν να συμμετέχουν στο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το ξέρω ότι δεν μπορείτε να εμποδίσετε του άλλου. Εσεί γιατί δεν θέλετε να μπείτε σε αυτό το θέμα. Θα βοηθούσε ε, ε, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε γιατί η ίδια η Προεδρία δεν συμμετέχει σε αυτό το γκρουπ για το φόρο ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Να σα πω γιατί είναι κακό για τα ταμεία τα συνταξιδοτικά, τα pension funds τα δικά μα, που είναι και πολλά. Είναι περίπου διπλάσια του ΟΕΚ, ο όγκο των συνταξιδοτικών ταμείων. Και αν είναι κάτι κακό των ταμείων αυτών που ε, αποτομιεύουν χρήματα για τους ηλικιωμένους, ε, τότε δεν είναι καλή ιδέα. Και το άλλο, το φόρος ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών προσκρούει σε ένα φόρο τραπεζικών τελών που χρησιμοποιούμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ωραία. Ο Πίρκουρ Ρόνεν Λέρνεν από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Thank you, Chair. Συγγνώμη, η κυρία Ρόνεν. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Βίμπες, με χαρά άκουσα τόσα είπατε για τη φορολογία. Οι απαντήσεις σας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φωτίζουν πάρα πολύ τα θέματα αυτά που είναι τόσο περίπλοκα και που χρειαζόταν τόσο να φωτιστούν. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω ε, ένα παράδειγμα διασυνοριακής ε, φοροαποφυγή. Ε, η Καρούνα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη Φιλανδία που ε, ε, ε, μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα. Το 2014 50 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στη Φιλανδία και επληρώσε μόλις 1,6%. 800.000 ευρώ για να είμαστε ακριβείς. Πώς είναι δυνατόν μπορεί να αναρωτηθείτε. Ποιο ήταν το τέχνασμα και αρκετά απλό. Ο μήλος ο Φιλανδικός έκανε ενδομιλικικά δάνεια προς την Ολλανδία, τάξιους εκατομμυρίων, που διάβρωσαν τα κέρδη της Καρούνα στη Φιλανδία και αυτές οι ενδομιλικές συναλλαγές επηρέασαν ε, και τα φορολογικά έσοδα της χώρας. Σε σχέση λοιπόν με το συγκεκριμένο παράδειγμα θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς είναι δυνατό και πώς προτίθεται η Ολλανδική Προεδρία να αντιμετωπίσει τέτοια φοροαποφυγή και να προλάβει και νέες περιπτώσεις ε, τύπου καρόνα για να μην ξανασυμβούν. Και επίσης, οι προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα αποδώσουν, δηλαδή θα είναι πιο δύσκολο κάτι τέτοιο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργός. Δεν θα σχολιάσω με μονομένες επιχειρήσεις τις οποίες δεν γνωρίζω. Αλλά να πω ότι αν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι τα κέρδη μιας επιχείρησης εγκαταλείπουν την χώρα και αυτό δεν είναι σωστό, τότε είναι σε θέση συγκεκριμένη χώρα να ζητήσει τη φορολογία μέσω των μέτρων αντικαταχρηστικής φορολογίας. Δηλαδή, η χώρα στην οποία έχει τη βασική έδρα η επιχείρηση αποφασίζει ποιο τμήμα των κερδών θα φορολογηθούν επί τόπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εσείς έχετε ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν ότι θα πρέπει να φορολογούνται τα κέρδη εκεί που δημιουργείται η αξία και αν η αξία δημιουργείται στη Φιλανδία θα πρέπει να φορολογηθεί στη Φιλανδία και δεν έχει καμία σχέση με άλλες χώρες, είτε είναι η Ολλανδία είτε η αδίποτε άλλη στην οποία ταξιδεύουν τα κέρδη. Η φιλανδική κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να φορολογήσει στο επίπεδο το οποίο θεωρεί σωστό. Τώρα πώς θα προλάβουμε τέτοια φαινόμενα. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φορολογικών συστημάτων και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές αυτές και με μέσα κατά των καταχρήσεων να διασφαλίσουμε έτσι ώστε μια σκοπούμενη τέτοιου είδους φοροαποφυγή να μην συμβεί. Υποθέτω ότι είναι μια τέτοια περίπτωση, δεν το ξέρω, επαναλαμβάνω. Πάντως το θέμα ακριβώς που συζητάμε είναι γεμάτο από τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό θέλουμε να αντιμετωπιστεί και θέλουμε η φορολογία να πληρώνεται εκεί όπου παράγεται η αξία. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις γύρω από τα φορολογικά, αλλά πάνω σε αυτή την αρχή οι περισσότεροι συμφωνούν απολύτως ότι θα πληρώνεται ο φόρος εκεί που δημιουργείται η αξία και ό,τι κάνουμε έχει σαν βασικό στόχο το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τώρα την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει σαν παράδειγμα ένα τμήμα του πακέτου το οποίο έχει ε, καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλαμβάνει και περιορισμούς στη μείωση των επιτοκίων έτσι ώστε επαναλαμβάνω να πληρώνεται ο φόρος εκεί που παράγεται η αξία. Λοιπόν, ίσως να υπάρχει θέμα, αλλά όπως σας είπα δεν γνωρίζω την υπόθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω. Πρώτον, σε σχέση με την ομάδα εργασίας... Εδώ μπροστά, εδώ μπροστά σας είμαι. Δεν μπορούσα. Πιο κοντά δεν γίνεται. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση σε σχέση με την Επιτροπή Κώδικα Διοντολογίας, COC του Συμβουλίου, σε σχέση με την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι πρόσφατα, 2 Φεβρουαρίου, εγκρίθηκε μια απόφαση αλλά για τις εξερχόμενες πληρωμές ε, δεν ελήφθη καμία απόφαση, δεν συζητήθηκε το ζήτημα. Αντίθετα με αυτά που είχαν αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας το φθινόπωρο που μας πέρασε. Εξερχόμενες πληρωμές λοιπόν, outbound payments, ε, δεν ε, ασχολείται η Ολλανδική Προεδρία με αυτό το ζήτημα. Γιατί εγκαταλείψατε το ζήτημα και διεθνώς έχετε ε, αυτή τη φήμη ότι είσαστε εξαιρετική θύρα εξόδου χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στη φορολογική σας νομοθεσία. Ε, χωρίς λοιπόν να γίνεται καταλογισμό σε κανένα προπολογισμό διαφεύγει το χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ε, σε σχέση τώρα με τα διάφορα φορολογικά καθεστώτα, των κρατών μελών. Εάν δεν υπήρχαν διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, δεν θα υπήρχε λόγο ύπαρξη για την τάξη 2. Και εσεί είσαστε φορολογικό παράδεισο στην Ολλανδία. Χιλιάδε επιχειρήσει έχουν τι οικονομικές δραστηριότητες τους στα επιμέρους κράτη-μέλη, όμως του φόρους τους πληρώνουν στην Ολλανδία, όπου έχουν μια, ε, ε, ένα γραμματοκιβώτιο. Είναι κάτι πλασματικές αυτές οι εταιρείες. Αυτά, αυτό είναι το σύστημα που ακολουθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και έτσι πολύ απλά δεν καταβάλλεται φόρος στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, αλλά καταβάλλεται σε άλλες χώρες, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δική σας. Μας μιλήσατε για το φορολογικό ανταγωνισμό και για το φορολογικό dumping και την φοροδιαφυγή, διότι ε, ξέρουμε ότι έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να μας δίνει μαθήματα στην Πορτογαλία και να μας κάνει κηρύγματα σε σχέση με πώς πρέπει να παρουσιάζουμε τα δημόσια οικονομικά μας. Ε, να σας πούμε και εμείς λοιπόν ότι δεν σας ανήκουν αυτοί οι φόροι που εισπράτεται. Ε, πώς θα αναλάβετε λοιπόν αυτή την ευθύνη σας, εάν γενικευτεί αυτό το φαινόμενο της Ολλανδίας, ε, θα υπάρχει πολύ πλευρό φορολογικό dumping και τελικά δεν θα είναι πλέον βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Και κλείνω με πολύ, ε, ένα πολύ απλό ερώτημα. Είπατε δεν θέλετε να αποφανθείτε, αλλά είναι πολύ απλό το ερώτημα. Με όλα αυτά ως δεδομένα, θεωρείτε δίκαιο να οικειοποιήσετε φορολογικά έσοδα που δεν σας αναλογούν. Ε, με το χαμηλό εταιρικό φόρο, τόσο χαμηλό συντελεστή που φτάνει και σε μηδενικά επίπεδα. Και ποια είναι η λειτουργία του κράτους λοιπόν ε, σε αυτά τα κράτη-μέλη όπως το δικό σας όπου παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστούμε. Ο υπουργό. Σας ευχαριστώ και για την ερώτηση. Μου είπατε γιατί βγάλαμε από την ημερήσια διάταξη τις εξερχόμενες πληρωμές. Μα δεν τις βγάλαμε. Είναι στο έγγραφο εργασίας του 2015, αυτό επεξεργαζόμαστε στο, στην Επιτροπή COC και είναι και στον οδικό χάρτη της Προεδρίας που λέει ότι μπορούμε να αρχίσουμε την άνοιξη της εργασίας για τις εξερχόμενες πληρώμες. Δεν το βγάλαμε από την μέση διάταξη το ζήτημα. Και μετά με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για το Ολλανδικό φορολογικό σύστημα. Δεν είναι ο σκοπός σημερινής μου επίσκεψης, σημερινής μου επίσκεψης αλλά θα ήθελα να σας δώσω κάποιο, κάποια απάντηση, επειδή είναι σοβαρό το ερώτημά σας. Λοιπόν, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι έχουμε εξαίρεση για τη συμμετοχή και δεν έχουμε φορολόγηση στην πηγή για, τα, ε, για τους στόχους και για τα δικαιώματα χρήσης. Για να ε, λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά και οι θηγατρικές να έχουν την ίδια θέση με τις τοπικές εταιρείες. Ε, θέλουμε να έχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τα έχουμε συμφωνήσει αυτά όλοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ολλανδία. Εφαρμόζουμε την ίδια αρχή, τίποτα περισσότερο, σε παγκόσμιο επίπεδο διότι η εσωτερική μας αγορά είναι μικρή χώρα, η Ολλανδία. Ε, ε, δύο βήματα να κάνετε έχετε πέρα διασχίσει τα σύνορα, η δική μας εσωτερική αγορά ε, εκλαμβάνουμε την εσωτερική αγορά όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ως παγκόσμια αγορά και όπως είπατε και εσείς από το 17ο αιώνα το ίδιο κάνουμε δεν έχουμε αλλάξει πρακτική κυρία Μάτια συμφωνώ παρόλα αυτά μαζί σας πως ε, κάποια ζητήματα που από κοινού όλοι εγκρίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που κάποιοι όπως εμείς ε, χρησιμοποιούνται παγκοσμίω ε, και που οδηγούν στη δυνατότητα για κάποιους να φοροαποφεύγουν, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς τρώμε και καταπίνουμε όλους τους φόρους και διότι η βασική αρχή για μας είναι ότι αν δεν υπάρχει προσθέμενη αξία δεν ε, φορολογείται κάτι. Οπότε δεν ισχύει αυτό για τις πορτογαλικές εταιρείε και θα σας δώσω και μια απάντηση όπως και ε, προ λίγων λεπτών στο συνάδελφο. Εάν η Πορτογαλία θεωρεί ότι αυτές, αυτοί οι φοροί κανονικά θα έπρεπε να καταβληθούν στην Πορτογαλία διότι η προσθέμενη αξία διαπιστώνεται στην πορτογαλική επικράτεια, τότε μπορεί να τους εισπράξει τους φόρους. Εμείς δεν είμαστε κατά, διότι δεν μας αναλογούν αυτοί οι φόροι. Η χώρα στην οποία κατευθύνονται οι φόροι μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά. Όμως ε, το θέμα είναι ότι οι πορτογαλικές αρχές πρέπει να αποφασίσουν ε, να ε, προβούν στη φορολόγηση αυτών των προϊόντων όπου παρατηρείται προσθέμενη αξία. Πρόεδρος, για να μην παρατείνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας άφησα άλλα δύο λεπτά γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Η κυρία Ματίας, ε, ε έχετε, είσαστε στην κυβέρνηση πλέον, οπότε να πάτε να τα πείτε στον Υπουργό Οικονομικών σας, ε, να του, το προτείνετε αυτό. Ερνέστ Ουρτασούν, στα πράσινο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Εδώ είμαι, Υπουργέ. Uh, Πρώτον, για τους κανόνες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, κάποια κράτη-μέλη, κάποια άλλοι δεν μπορούν. Γι' αυτά είναι τα tax rulings. Και έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση υπόψη μας σε απόφαση για τη Starbucks της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποφασίσατε να κάνετε έφεση. Ε, καταλαβαίνετε ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας δεν ε, καλοδέχονται αυτό και θεωρείτε πολύ οικοδομητική αυτή τη στάση σας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγή. Πρώτη ερώτηση αυτή. Άλλες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την έκθεση για την IKEA ε, που δημοσίευσε η δική μου ομάδα πριν από λίγε μέρες. Ε, και ξέρουμε ότι ε, είναι τα προβλήματα γνωστά της εταιρεία ε, σε πλήρη εχεμήθεια και μυστικότητα. Πολλά αυτά τα λέει και πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση που σας έκανε ο κύριος ε, Μπαγιέ. Ε, βλέπουμε τον κίνδυνο να σπάσει στα δύο την πρόταση το Συμβούλιο και να μην ερευνήσει το ένα σκέλος. Ε, δεσμεύεστε ως Προεδρία, γιατί απαντήσατε κάπως αόριστα, έτσι ώστε το πακέτο αυτό να παραμείνει ένα, μια νέα δέσμη και να αποφύγουμε να σπάσει τα δύο και να μην ασχοληθούμε καθόλου με το ένα. Και τελευταία τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με την ελάχιστη φορολόγηση ε, των ε, δικαιωμάτων και επιτυχίων που συζητάει τώρα η Ευρωπαϊκή, το Συμβούλιο μάλλον στην αντίστοιχη οδηγία. Οι κάτω χώρες έχουν ένα ευρύ δίκτυο ε, διπλών ε, μορφών φορολόγησης που επιτρέπει σε ε, εταιρείε να φοροδιαφεύγουν και τα δικαιώματα τα φορολογείται με 5% ενώ ο φόρος επιχειρήσεων είναι 25% σε κάποιες περιπτώσεις. Έχετε προτείνει ένα ελάχιστο 10% για τα δικαιώματα και αν ναι, για ποιο λόγο τόσο χαμηλό φορολογικό συντελεστή. και θέλω να ρωτήσω πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε ε, την πρότασή σας να εξαιρείτε από το 10% του κατώτατου συντελεστή καινοτομία και ε, ε, οι ευνοϊκές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα patent boxes. Γιατί εμείς έχουμε, φορολογι... Ε, έχουμε μάλλον στην Επιτροπή μας εδώ κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι πρόσφορο το Ολλανδικό μοντέλο να ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο Υπουργέ για να απαντήσετε. Um, Ευχαριστώ κύριε Ούτασο. Πράγματι εμείς υπογράψαμε έτσι ώστε να ανακληθεί η απόφαση της Επιτροπής για τη Starbucks. Και επανέρχομαι σε κάτι το οποίο είχα πει και στο παρελθόν. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να φορολογούνται τα κέρδη εκεί όπου παράγεται η συγκεκριμένη αξία. Αν κάτι δεν πάει καλά στο Ολλανδικό σύστημα, με μεγάλη ευχαρίστηση θα το επισκευάσουμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας υποχρέωσε να φορολογήσουμε κέρδη ενώ η αξία δεν είχε ε, παραχθεί στην Ολλανδία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε χρησιμοποιήσει ένα ίδιο κριτήριο για τον υπολογισμό των κερδών το οποίο δεν αντικατοπτρίζει τους κανονισμούς του πλαισίου ΩΣΑ. Εμάς μας ικανοποιούσε το πλαίσιο ΩΣΑ, το πλαίσιο ΜΠΕΠΣ. Το πλαίσιο ΜΠΕΠΣ ήταν σαφές, ήταν λεπτομερές και σε επίπεδο τεχνικό ιδιαίτερο επαρκές. Εμείς έχουμε αναλάβει πλήρως την υποχρέωση να εφαρμόσουμε πλήρως το πακέτο του ΟΣΑ για τη μεταφορά ή τη μεταβίβαση μάλλον των τιμών η Ολλανδική κυβέρνηση λοιπόν ή το ευτυχής ή το σύμφωνη με την πρόταση BEPS του ΟΣΑ είναι κάτι το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα και δημιουργεί ένα ομοιογενές παγκόσμιο σύστημα. Αλλά ήρθε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δεν ήταν συμβατή σε καμία περίπτωση με αυτή τη λογική. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι παραβιάστηκε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κανονισμός ΩΣΑ. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε εμείς να ζητήσουμε την νομική βεβαιότητα. Εφόσον ο ΩΣΑ λέγει στον κόσμο ότι θα πρέπει να κάνουμε το Α και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Β, τότε αυτό δημιουργεί ένα επίπεδο αβεβαιότητας το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Για τη δεύτερη ανησυχία σας κύριε Ούρτασον σχετικά um, the, um, με την ADAP, την πρόταση ADAP. Uh, λοιπόν, σχετικά με το ATAP, θα ξεκινήσουμε με το μεμονωμένο πακέτο και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο του πακέτου και να το ολοκληρώσουμε. Στο τέλος όμως κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα. Εμείς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να καταλήξουμε στις περισσότερες από τις προτάσεις μέχρι τώρα. Yeah, και τώρα τι γίνεται με τα innovation boxes, με τις ευρεσιτεχνίες την καινοτομία και τι γίνεται επίσης ε, με τις οφειλές και τα επιτόκια. Είπα στην εισαγωγή μου ότι αυτός είναι ένας τομέας στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το IRD και προσπαθούμε να συζητήσουμε μήπως και καταλήξουμε κάπου. Σας ευχαριστώ. Η Ατζέα έχει το λόγο για το FDD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον Υπουργό. Ήρθατε εδώ πραγματικά να κάνετε μία μορφή χαρακήρη στην Επιτροπή. Είναι μία από τις λίγες φορές που τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερος φιλόδοξο θα έλεγα και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι λόγος ε, συγκυρίας, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας πλέον. Και το άλλο είναι ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κρατη που είναι πολύ δύσκολα συμβιβάσιμες. Από την άλλη θα ήθελα να εκφράσω την ευαρεσκιά μου για το ότι η Ολλανδία είναι αυτή που θα καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις. Έχετε λειτουργήσει στον τομέα της βελτιστοποίησης των φορολογικών εσόδων, έχετε καταστήσει τη μέθοδο αυτή ιδιαίτερως ελκυστική περισσότερο από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, ποια έρευνα είναι αυτή που λέει ότι στην Ολλανδία υπάρχουν 12.000 επιχειρήσεις ε, γραμματοκιβώτια ε, για 12 δις ε, εισπράξεις φόρων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο μεγάλη αξία επιχειρηματική και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απλές ταχυδρομικές διευθύνσεις και δεν θα υπογραμμίσω το ότι ανάμεσα σε αυτές τις 12.000 επιχειρήσεις γραμματοκιβώτια υπάρχουν 80 από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος παγκοσμίως. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν εκπλήσωμε βέβαια, γιατί από τη μία εσείς επιβάλλετε τη λιτότητα στα δημοσιονομικά των κρατών, αλλά επιτρέπετε στις ίδιες τις χώρες να κάνουν ανταγωνισμό προς τα κάτω, η φορολογία των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών και των μεγάλων βιομηχανιών. Γι' αυτό πρέπει να περικόπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο κοινή ωφέλεια και δυστυχώς να αυξάνεται ο τζίρος, ο κύκλος εργασιών των μεγάλων επιχειρήσεων. Βλέπω εγώ ποια είναι τα αποτελέσματα τα εξαιρετικά των οικονομικών σας αποφάσεων. Επανέρχομαι στα λεγόμενα ούρτα σου για την ε, γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επιχείρηση Starbucks, όπου η Ολλανδία έχει ε, καταθέσει την αντίρρησή της και ε, θεωρήθηκε ότι η Ολλανδία χρησιμοποίησε κρατικές επιδοτήσεις εις βάρος των, των κανόνων που ισχύουν. Δεν είναι παράδοξο τελικά που οι ίδιες χώρες που κάνουν ειδικέ φορολογικές συμφωνίες και οι οποίες στην ουσία πληρώνουν τα πρόστιμα τα οποία τους καταλογίζονται που δεν είναι τίποτα βέβαια σε σχέση με τα πραγματικά κέρδη και σε σχέση με τη φορολογική ζημία την οποία προκαλείται σε άλλες χώρες και για το λεγόμενο switch over και η, Ένωση Ολλανδών νομομαθών στον τομέα της φορολογίας έχει εκφράσει επιφυλάξεις. Σας ευχαριστώ, ζητώ από τους συναδέλφους να μην θέτουν ε, ε, πάρα πολύ μακρόχρονες ερωτήσεις. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Δεν άκουσα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις να είμαι ειλικρινής για να μπορέσω να απαντήσω σε όλες αυτές. Η ερώτηση θα, πρέπει, θα μπορούσε να απαντηθεί είτε σε δύο δευτερόλεπτα είτε σε δύο ώρες. Απλά πρέπει να κάνω μια επιλογή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι παράδοξο αυτό το οποίο είπατε. Η καλύτερη απάντηση την οποία μπορώ να δώσω στην κυρία Άτζεα είναι να έρθει στην Ολλανδία και να πιστεί ότι στην Ολλανδία δεν υπάρχουν μόνο τα φορολογικά έσοδα. Να τη πω επίσης ότι οι ροές οι χρηματικές είναι μερικές φορές κάτι το εντελώς διαφορετικό από την αξία. Δεν αποδίδουν και τόσο για την Ολλανδία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Από την ΕΝΕΦ. E ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να μου απαντήσετε, γιατί έκανα συγκεκριμένε ερωτήσει, πάρα πολύ συγκεκριμένε. Είναι και ένα είδο στοιχειώδου σεβασμού να απαντήσετε σε κάποιε ερωτήσει από αυτέ που έκανα. Bien. Euh, le ministre... Καλώς. Απάντησε ο Υπουργός. Ο κύριος Άνεμανς από την ομάδα ΕΝΕΦ. Χωρίς μικρόφωνο. Υπουργέ, έχετε τίποτα να προσθέσετε για 30 δεύτερα. Μία από τις ερωτήσεις που έφτασε προς το τέλος ε, δεν ξέρω αν ήταν επίσημη ερώτηση, ε, τι πιστεύουμε ως χώρα για τη ρήτρα switch over. Αυτό δεν ήταν μεταξύ των ερωτήσεων. Κάπου το προσθέσατε στο τέλος και το κόψετε για λόγους χρονικούς. Νομίζω ότι είναι άκρος αντιπαραγωγικό, αν ε, οι Ολλανδοί τώρα αρχίζουν να έχουν γνώμες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας τους. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θεωρεί σημαντικό και ο Γιουρούν Ντάισελμπλουμ, πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και υπουργό οικονομικών μα. και ο ίδιο ο πρωθυπουργό μα θεωρούν πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μα και να είμαστε ένα έντιμο διαμεσολαβητή ω Προεδρία. Και δεν βοηθάει να έχουμε διάφορε απόψει ω Προεδρία για διάφορα θέματα. Ειλικρινά, θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητη Προεδρία, ε, ε, αμερόληπτη και ε, διαμεσολαβητής. Αυτό είναι η Προεδρία και όχι να έχουμε διάφορες απόψει για διάφορα θέματα. Αυτό το εξάμεινο θα προσπαθούμε να ε, καταλήγουμε σε συμφωνίες για όσο γίνεται περισσότερες από τις προτάσεις που μας απασχολούν. Ο κύριος Άνεμαν από την Ευρώπη τη ελευθερία και των Εθνών. Ευχαριστώ. Ε, Χαίρομαι που έχουμε ένα ε, δεξιό φιλελεύθερο από την Ολλανδία, γιατί συνήθως βλέπουμε τον σοσιαλιστή Ντάισελμπλουμ και ε, ευρωπαϊστή και φίλο του ευρώ. Άκουσα τη συζήτηση και τώρα η Ολλανδία λέει είναι μια χώρα που έχει μπει στην περίπλοκη αυτή ε, κατασκευή έχουμε το Double Irish, τώρα έχουμε και το Dutch Sandwich. Όλοι αυτοί οι ορισμοί δεν είναι ουρανοκατέβατοι και δεν είναι και τυχαίοι. Και κανονικά θα πρέπει να απαντήσετε για την αξιοπιστία της Ολλανδίας, ε, των κάτω χωρών. Έχω μια ειδική ερώτηση. Διάβασα από τον Ολλανδικό τύπο, κυκλοφορούν εκεί κάτι φήμες, ότι ο κύριος Ποροσέγκο, ο Ουκρανός, μέσω ενός κατασκευάσματος στην Ολλανδία και στην Κύπρο, 1,7 δισεκατομμύρια έχει βγάλει από την Ουκρανία. Μέσα από το καρουσέλ του Άμστερνταμ που κυκλοφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια, ε, άλλος ε, ορισμός ε, από αυτόν τον κόσμο, λίγο μυστήριο μου φαίνεται αυτό ως κατασκευή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλάει για 11 δισεκατομμύρια που έχει στείλει στην Ουκρανία, σε μια χώρα που δεν καταβάλλονται οι φόροι και φεύγει ο πρόεδρος με ένα Λονδικό κατασκεύασμα. Τα έχετε μάθει αυτά, τις φήμες αυτές τις ακούτε, τις ξέρετε, παίρνετε αποστάσεις και με ποιο τρόπο. Προσωπικά είστε υπέρμαχος του γεγονότος ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και στο δημοψήφισμα που επίκειται για την Ουκρανία στην Ολλανδία θα παίξει ρόλο αυτό. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός. Well, unfortunately I Δυστυχώς δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένες περιπτώσεις και εδώ δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά δεν ξέρω καν περί τίνος πρόκειται. Προφανώς γενικά όταν υπάρχει ένα στοιχείο απάτης και όπου υπάρχει απάτη και αν υπάρχει απάτη θα πρέπει να διώκονται οι απαταιώνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που δεν βρίσκει εφαρμογή δεν το γνωρίζω. Μα τα, κατά την άποψή σας λέει ο κύριος Άνεμας δεν ξέρετε ότι έχει θηρίδα και διεύθυνση ε, ο κύριος Ποροσέγκο στην Ολλανδία. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ, πρώτη φορά το ακούτε. Διαβάζω και εγώ τον τύπο, αλλά δεν σημαίνει ότι γνωρίζω την υπόθεση. Και ε, στο Ολλανδικό Δίκαιο υπάρχει μια ρήτρα που λέγει ότι ο Υφυπουργό ε, Φορολογίας ούτε ενημερώνεται για με μονομένους φορολογούμενους ούτε έχει καμία σχέση. Και φαίνεται περίεργο ότι υπάρχουν χώρες, κυρίως εκτός της Ευρώπης, όπου με μονομένοι υπουργοί και υφυπουργοί υποτίθεται ότι ενέχονται σε μονομένε περιπτώσεις και οι χώρες αυτές δεν είναι καλύτερες από την Ολλανδία. Εγώ επιμένω σε αυτό ότι ε, προσωπικά εγώ δεν ασχολούμαι με συγκεκριμένες υποθέσεις, είναι καλύτερα γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα δυστυχήματα ε, και ε, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, λέει ο κύριος Άνεμας. Αλλά θα γίνει δημόσια συζήτηση για ένα δημοψήφισμα που είναι τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσατε να κάνετε κάποια εξαίρεση στην περίπτωση αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ναι. Ε, καλά το καταλάβατε, λέει ο Υπουργό. Σα προτείνω το εξή να διαβάσετε γραπτός το ερώτημά σας, ούτως ώστε να λάβετε και ε, γραπτή απάντηση. Ευχαριστώ σίγουρα, Πρόεδρε, θα ανταποκριθώ σε αυτή την υπόδειξη και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Έστερ Ντελάνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω και να δούμε όλο το κλίμα το επενδυτικό, όχι μόνο στη δική μας παρτίδα, ε, βέβαια εγώ είμαι κόμμα της αντιπολίτευσης τώρα και μπορεί να έχω τελείως διαφορετικό ρόλο διακριτό από άλλους ευρωβουλευτές. Ανεξάρτητα από αυτό πώς έχει το επενδυτικό κλίμα. Ακούω λίγα πράγματα για να μην μιλήσω για την Ευρώπη καθόλου και τι γίνεται εκεί ως επενδύσεις. Τι επιρροή έχει το φορολογικό καθεστώς ε, στο συλλογικό επενδυτικό κλίμα. Το έχετε μελετήσει αυτό, το έχετε ψάξει και τα συμπεράσματα, ποια συμπεράσματα βγάζετε από ε, αυτές τις έρευνες και τις μελέτες ε, που κάνετε ή που έχετε στη διάθεσή σας και στα πλαίσια της συζήτησης που κάνουμε σήμερα μεταξύ μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργό. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό το ζήτημα. Είπα στην εισαγωγή μου θέλουμε να επικρατήσει φορολογική δικαιοσύνη και να είναι δίκαιες οι σφορές ε, φορολογικές φορές ε, στα δημόσια οικονομικά. Ταυτόχρονα όμως ε, θέλουμε εν γέννη στην Ευρώπη να επικρατήσει ένα ευνοϊκότερο επιχειρηματικό κλίμα. Είναι λοιπόν σημαντικό να προωθήσουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Και γι' αυτό τα... είναι τόσο χρήσιμο το BEPS σε παγκόσμιο επίπεδο. δεκαετίες ολόκληρες ε, αναρωτιόμασταν ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση και αν προκύπτει η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή από διαφορές των εθνικών συστημάτων, τότε ποιος κάνει την πρώτη κίνηση. Και το σύστημα BEPS ε, αυτή την ομορφιά έχει ότι κάνουμε ε, από κοινού το πρώτο βήμα. Και γι' αυτό ε, σε διεθνές επίπεδο είναι ισότιμη όρια ανταγωνισμού. Τι είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη να ακολουθήσουμε κατά, ε, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τις, τα πορίσματα και τις συστάσεις ε, του ΩΣΑ με τον ίδιο περίπου ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό θα είχε ιδιαίτερη σημασία. Και γι' αυτό και σε αυτό μας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να κάνουμε βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα με βήματα που γίνονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Σημαντικά τα φορολογικά, αλλά δεν είναι και τα μόνα ζητήματα. Ξέρουμε ότι η ασφάλεια, οι καλές καιρικέ συνθήκες, έχουν επίσης ε, ε, ειδικό βάρος. Ε, δεν διαλέγει κάποιος μόνο βάσει του, του φορολογικού συστήματος. Υπάρχουν χώρες με ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που παρόλα αυτά παραμένουν μη ελκυστικές λόγω του κακού επιχειρηματικού κλίματος. Χρειάζεται ένα συνολικό μίξε. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στη φορολογική πολιτική. Κυρία Τζέα, γι' αυτό σας είπα να έρθετε, να έρχεστε μάλλον, να επισκέφτεστε την Ολλανδία, να βλέπετε ειδήσω όμως τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε. Ε, Ρέμουρ Χαουρέγγι. Μα έχω άλλο ένα λεπτό. Εκτός σε μικροφόνο ο Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας μιλήσω για το ρόλο σας ως την Ολλανδική Προεδρία ε, σε αυτή την κοινωνική αναταραχή και το συναγερμό που ζει ο κόσμος για θέματα φορολογικά στην Ευρώπη. Πρέπει να καταλάβετε ότι πολλοί από τους συναδέλφους μου εκφράζουν μια αμφιβολία όχι μόνο για το ποια μπορεί να είναι η φορολογική πολιτική στην Ολλανδία, αλλά γιατί εδώ και πολλά χρόνια η χώρα σας σε αυτά τα θέματα του φορολογικού συντονισμού έχει δραματίσει ένα ρόλο που μας κάνει να αμφιβάλλουμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχετε ασπαστεί τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί. Αλλά επειδή διάβασα τα πρακτικά ε, του, της ομάδας για την, τον κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου και είδα ε, τόσες ευνοϊκές ολλανδικές θέσεις στη, χαμηλή φορολογία παντού, θεωρώντας ότι δεν είναι πρόβλημα, ότι δεν είναι μυστήριο ε, υπερασπίζεστε τόσο πολύ το απόρριτο και είστε τόσο αντίθετοι στο ίδιο το μέλλον της ομάδας ε, για τον κώδικα διοντολογίας που εδώ στο Κοινοβούλιο ε, υπάρχει ζήτηση να παίξετε ένα ρόλο, πώς να το πω, διακριτό από το μέχρι τώρα και τη σταδιαδρομή και την πορεία της χώρας σας. Τώρα, αν πέσατε από το άλογο και ασπαστήκατε τον συντονισμό, θαυμάσια, αλλά σαν τον Απόστολο Παύλο, ξέρω εγώ από Σαούλ. Ε, καλά τα λέτε εδώ, αλλά εγώ έχω διαβάσει και τα πρακτικά και ξέρω ποια είναι η Ολλανδική θέση για αυτό το θέμα και θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύετε, έχει ρόλο να παίξει στο συντονισμό και στην εναρμόνιση για τα φορολογικά στι τελευταίε οδηγίε ή όχι γιατί το Συμβούλιο προσπαθεί να αποφύγει να δώσει ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πρωταγωνιστεί σε όλη αυτή την προσπάθεια συντονισμού, εναρμόνισης κλπ. στα φορολογικά θέματα. Ακόμα και στον ίδιο το κώδικα διοντολογίας. Και δεύτερη ερώτηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπατε για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Βέβαια μας είπε και ο Πρόεδρος ότι δεν είναι αντικείμενο της δικής μας ε, Επιτροπής. Να σας ρωτήσω, υπάρχει μεγάλη απάτη στη διασυνοριακό ΦΠΑ. Μπορείτε μια τάξη μεγέθους να μας δώσετε. Ένα ποσοστό φορολογικής απάτης στο ΦΠΑ στην Ευρώπη στις διασυνοριακές συναλλαγές. Θα ήταν πάρα πολύ ε, χρήσιμο να το ξέρουμε και σημαντικό για μας. Ευχαριστώ πολύ ο Υπουργός. Um, well, in general, one I think the... Νομίζω ότι τέθηκαν και πολλές έμεσες ερωτήσεις. Μία από αυτές ζητά τη γνώμη μου σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά φορολογικής επιβολής στα πλαίσια του φορολογικού ανταγωνισμού. Αυτή είναι η ερώτησή σας. Εγώ είπα στην εισαγωγή μου ότι δεν θέλουμε εμείς να συζητήσουμε συγκεκριμένα συγκεκριμένες Ολλανδικές θέσεις. Θέλουμε γενικά οι προτάσεις που είναι υποσυζήτηση να γίνουν τελικά δεκτές. Και νομίζω ότι η ταχύτητα με την οποία προσπαθούμε να το πετύχουμε είναι ιδιαίτερο υψηλή. Γενικά πιστεύω επίσης ότι το θέμα αυτό είναι έμπλεο προτάσεων για την αποφυγή της φοροαποφυγής και επίσης να σταματήσουν να δημιουργούνται κάποια σχήματα τα οποία οδηγούν σε φορολογικά έσοδα να διαφεύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα επίπεδα φορολογίας πρέπει να οι συντελεστές οι φορολογικοί πρέπει να εναρμονιστούν. Ξέρετε ότι ανάμεσα και στις διάφορες χώρες ε, στο ΕΚΟΦΗΝ Υπάρχει σαφέστατη πεποίθηση ότι το θέμα των φορολογικών συντελεστών είναι εθνικό θέμα. Ο φορολογικός ανταγωνισμός υπάρχει, δεν είναι θέμα απλά να πούμε ότι είναι τμήμα της ζωής, αλλά υπάρχει και κάτι εξυπηρετεί. Και ταυτόχρονα η μη ε, σκοπούμενη, ή μάλλον η σκοπούμενη φοροαποφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα φορολογικά συστήματα πρέπει να εναρμονιστούν. Ίσως να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να συμφωνούμε σε μέτρα εναντίον των καταχρήσεων. Δεν είναι η εναρμόνιση το μοναδικό μέσο για να μην διαφεύγουν τα φορολογική έσοδα. Τώρα διαμεθοριακές απώλειες και απάτες στον τομέα του ΦΠΑ. <coughs> δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς αυτά τα οποία δεν μπορεί να γνωρίζει. Οι εκτιμήσεις είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους. Κάποιες αναφέρονται σε εκατοδείς δις απώλειες εσόδων. Αλλά πάντως γενικά μιλάμε για απάτες, για κλοπή δηλαδή, για μια ποινικά κολάσιμη δραστηριότητα δεν μιλάμε για σχήματα, μιλάμε για κλέφτες οι οποίοι κλέβουν από το κράτος τα είσοδά του και κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα ήδη στην διάθεσή μας και είμαι διατεθειμένος να πιέσω, να πείσω τους συναδέλφους στο Συμβούλιο ότι κάτι πρέπει να γίνει, να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε και να δούμε ποιοι είναι οι απαταιώνες. Εμείς έχουμε διάφορα μέσα, αναπτύξει ένα τέτοιο μέσο έχουμε και εμείς στην Ολλανδία και το χρησιμοποιούμε με μια κάποια επιτυχία λέγω και θα θέλαμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Η Εστέρ την οποία διέκοψα προηγουμένως δυστυχώς. Έχω και άλλη ερώτηση για την κοινή ενωπημένη βάση φορολόγησης. Θα το πω στα Ολλανδικά. Ε, όταν η ρήτρα κατανομής είναι για τον κοινό ενοποιημένο, κοινή ενωπημένη βάση για τον εταιρικό φόρο. Ε, υπάρχουν διαφορές στις οικονομίες των διαφόρων κρατών μελών, έτσι, προϊόντα, υπηρεσίες κτλ. Ποιος θα πρέπει να είναι σχετική αυτή η κλίδα για την κατανομή ανάλογα ε, με τον πληθυσμό και όχι απόλυτη, όχι απλώς να κοιτάμε για την εργασία που δημιουργεί κάθε, ή τον κύκλο εργασιών που έχει κάθε επιχείρηση. Γενικά εδώ ε, θέλουμε ένα κοινό ενοποιημένο σύστημα, κοινή ενοποιημένη βάση, όχι απλώς μια κοινή βάση, αλλά και το C, το consolidate μας ενδιαφέρει η ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Και τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε μια λύση, δεδομένου ότι απαιτείται ομοφωνία. Ευχαριστώ, υπουργό. Um, well, ναι, λίγο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό, διότι η πρώτη πρόταση, η CCCTB, ενοποιημένη βάση, δεν έτυχε θετικής ε, υποδοχής από την Ολλανδική Βουλή, όπως τα ξέρετε ενδεχομένως, ήταν μάλλον ε, αρνητική στάση και το ίδιο η στάση της κυβέρνησης. Γιατί, διότι σε αυτή την κλίδα ανακατανομής του κερδών, διότι περί αυτού πρόκειται, λέμε ουσιαστικά ε, ότι ε, αποφασίζει η κλίδα που θα επιβληθεί η φορολόγηση και όχι ο τόπος στον οποίο υπάρχει κάποια παραγωγή. Ε, όμως αναμένεται άλλη πρόταση, την οποία δεν έχω δει ακόμη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι, δεν είναι παραγωγικό λοιπόν να αρχίζω εγώ τώρα να αναφέρομαι σε απαιτήσει, προαπαιτήσει που θα είχαμε για μια τέτοια ανύπαρκτη ουσιαστικά πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σχολιάζω δηλαδή ε, αποφάσεις, ε, προτάσεις γνώμη που έχει εξαγγείλει η Επιτροπή αλλά που δεν υφίστανται ακόμη δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ. Υπερβάνω σπέρα. Ευχαριστώ. Θα τα πω στα αγγλικά. Διότι καμιά φορά λέτε δεν καταλαβαίνετε τα γαλλικά, θέλω να είμαι σίγουρη, λοιπόν θα τα πω στα αγγλικά. Το σύστημα Starbucks ε, υπάρχει καταδικαστική απόφαση για τη χώρα σας ε, και δεν μπορείτε να αρνηθείτε την ε, υπηκότητά σας. Ναι, εκπροσωπείτε την Προεδρία αλλά και την Ολλανδία. Οπότε πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση της λειτουργίας στην Ολλανδία, να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις από την Ολλανδία για να αναβαθμίσετε λοιπόν το ευρωπαϊκό σύστημα. Έχοντας αυτά κατά νου, στο μέλλον τι θα κάνετε ώστε ε, να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ε, ε, για την οποία σας αποδόθηκαν ευθύνε για να καταστεί αδύνατο ένα τέτοιο φαινόμενο στο μέλλον. Γιατί CCTV είναι πλήρες το παράδεξο. Λέτε αφενός που δεν θέλετε να επιβάλλετε φορολογία εκεί που δεν παράγεται η προστιθέμενη αξία, όμως όταν μιλάτε για την κλίδα κατανομής είναι προφανές ότι κανείς δεν γνωρίζει που έχει παραχθεί η αξία. Δεν μπορείτε δηλαδή να λέτε ένα πράγμα και το αντίθετο του ταυτόχρονα και είπατε πως δεν έχει υποβάλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί εσείς ως Ολλανδός να μην ξέρετε τι θα ήταν το καλύτερο να συμβεί. Τρίτον, Θέλουμε το σύστημα του ΩΣΑ ή θέλουμε το σύστημα που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε ιδρυτική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι οφείλετε να υπερασπιστείτε το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσθέσει αξία στην πρόταση του ΩΣΑ μετά και την ερώτηση του συναδέλφου Μπαγιέ, δεν κρίνετε κι εσείς ότι χρειαζόμαστε ορισμό του TST διπλώμα ευρεσιτεχνίας. Είναι απαραίτητο αυτό. Και τέλος, ένα σχόλιο, ένα, αλλά μπορείτε να σχολιάσετε κι εσείς το σχόλιο μου. Είπατε πως η ελκυστικότητα ενός κράτους δεν συνδέεται αποκλειστικά με το φορολογικό σύστημα. Αχα. Οπότε για ποιο λόγο επηρεαστίζεστε αυτό το σύστημα που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό. Για σας ενώ σίγουρα θα είχατε και άλλα θέλγητρα για τους επενδυτές. Ευχαριστούμε αγαπητέ συναδελφέ. Ε, ο Υπουργός το έχει τον λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να, να ασχοληθώ με το πρώτο σας ερώτημα. Starbucks. Κυρία Μπερές, ότι υπονοείται Πώ είναι δύσκολο κανείς να έχει δύο διαφορετικά καπέλα, δύο διαφορετικέ ιδιότητε, δηλαδή να έχει τα ενία τη Προεδρία και ταυτόχρονα να λειτουργεί ε, αμερόληπτα ε, για την περίπτωση Starbucks. Μα εμείς δεν ε, επηρεάζουμε καθόλου την έκβαση τη υπόθεση. Είναι δικαστικό πλέον το ζήτημα. Δεν είναι στα χέρια μα ούτε και στα χέρια τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα σα καταδίκασε η Επιτροπή, λέει η κυρία Μπεριστά, κάνετε στο μέλλον για να μην ξανασυμβεί. Αυτό σα ρώτησα απάντηση. Να περιμένουμε την ε, απόφαση, να δούμε τι λέει και αν ε, υπάρχει πρόβλημα θα το φτιάξουμε. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα θα ακολουθήσουμε, έχουμε λάβει τη δέσμευση, ε, να ακολουθήσουμε τον ΠΕΠΣΕ για τη μεταβίβαση των κερδών και την φορολόγηση εκεί όπου δημιουργείται προσθέμενη αξία. Το έχουμε δηλώσει αυτό ήδη, δεν είναι γνωστό της πάσης την τώρα. αν ε, κάποια κέρδη ανήκουν σε μια χώρα και εκεί πρέπει να φορολογηθούν. Ποιο ήταν το κριτήριο μέχρι στιγμής, ε, η μεταβίβαση κερδών, ε, τιμών, συγγνώμη, the transfer pricing και οι κανόνες για τη μεταβίβαση τιμών έχουν εκπονηθεί πολλοί από τον ΩΣΑ έχουν ε, και διεθνή πρότυπα για τη μεταβίβαση των τιμών, ε, για να ξέρουμε ε, πού πρέπει να αποδοθεί κάθε κέρδος. Αυτά είναι τα παγκόσμια πρότυπα που ενέκρινε ο ΩΣΑ και αυτό διαφέρει από το θέμα της κοινή ενοποιημένης βάσης. Και για να περάσω και στο τρίτο ερώτημά σας, ναι, έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει ή να προσθέσει αξία όπως το θέσατε εσείς στην πρόταση του ΩΣΑ. Γι' αυτό έχουμε και την Επιτροπή, αλλιώς να την καταργήσουμε και να την εγκαταστήσουμε με τον ΩΣΑ. Βεβαίως ε, μπορεί να προσθέσει αξία η Επιτροπή και είναι δουλειά της Προεδρίας να το συζητήσουμε τα κράτη-μέλη και να καταλήξει σε μια συμφωνία για το μέγιστο δυνατό αριθμό προτάσεων της Επιτροπής και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Λέτε γιατί υπερασπίζομαι εγώ αυτό το σύστημα του patent box για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ε, δεν είχα την εντύπωση ότι το ΕΟ κάναμε αυτό, διότι υιοθετήσαμε και στον ΩΣΑ ε, και στην Επιτροπή Κώδικα Διοντολογίας έχουμε υιοθετήσει προσέγγιση έξω, οπότε αυτή την άγουσα θα ακολουθήσουμε και θα τροποποιήσουμε μόνο εάν χρειαστεί, δεν υπερασπιζόμαστε κάτι συγκεκριμένο. Αν υπάρχει κάποιο τελεσμένο, θα λειτουργήσουμε από αυτή τη βάση. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος της ακρόασης. Θα ήθελα να δώσω και πάλι τρία λεπτά σε κάθε συνεισηγητή για να, κάνουν, να βγάλουν κάποια συμπεράσματα από τη σημερινή συζήτηση. Κόφωτε Γέπε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε και Vibes ε, για τις απαντήσεις που μας δώσατε για το ρόλο της Προεδρίας αλλά και τις απαντήσεις που δώσατε ως εκπρόσωπος της Ολλανδικής Κυβέρνησης. Νομίζω ότι νομιμοποιούμαστε να θέτουμε τέτοια ερωτήματα εφόσον εκπροσωπείται εδώ η Ολλανδική κυβέρνηση και φυσικά γνωρίζοντας την κατάσταση στην Ολλανδία και τα βιώματα πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο ώστε για τον ανταγωνισμό να υπάρχουν ισότιμοι όροι και να μην υπάρχουν παράνομες κρατικές ενισχύσεις μέσα από φορολογικές διευκολύνσεις, όπως δηλαδή βλέπουμε σε διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να το αποκομίσετε από τη σημερινή συζήτηση. Πέραν αυτού, ήθελα να σας πω πως από πλευράς του Κοινοβουλίου και Τη Επιτροπής λέτε ότι εσείς είσαστε διαμεσολαβητή, συντονιστή, τέλος πάντων προσπαθείτε να διευκολύνετε την εξέβρεση συμβασμών. Καλό αυτό. Όμως ε, ταυτόχρονα να σημειώνετε τα μηνύματα που σας διαβάζουν ε, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και τις προτάσεις μας για την αποφυγή επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και τη φοροαποφυγή φοροδιαφυγή. Στην ε, έκθεση της ΤΑΞ 1 έχουμε πολλές τέτοιες συστάσεις ε, και θα σας ενθάρρυνα να τη διαβάσετε προσεκτικά. Το θέμα του συστήματος Patent Box ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι νομίζω πρόσφορο να λάβετε υπόψη αυτά που σας είπαμε. Προσβλέπουμε στην συνεργασία με τον Ολλανδική Προεδρία. Θέλω όμως να τονίσω ταυτόχρονα πως, όπως είπαμε και στην αρχή, Ας κάνουμε κάτι για αυτόν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό που μας οδηγεί όχι μόνο σε έναν όρου ανταγωνισμού αλλά και στο φαινόμενο ότι 30% μεγαλύτερο φορολογικό βάρος φέρουν οι μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με τις πολυεθνικές. Ε, και επίσης ε, ε, υπάρχει κλοπή φορολογικών εσόδων από κράτη-μέλη και αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα δαπανίσουμε για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για την κοινωνία Χρειαζόμαστε συνεργασία και γιατί το φορολογικό ανταγωνισμό Έχουμε συγκεκριμένε προθέσει εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο και το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ το ΕΡΕΡ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμη Υπουργέ, καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ανταλλαγή απόψεων εδώ με την Ολλανδική Προεδρία ανταλλαγή την οποία επιζητεί η Προεδρία σας, την οποία ποντάρουμε και εμείς την Προεδρία και ε, γι' αυτό το θέμα της αποφυγής ε, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Πιστεύω ότι θα κάνουμε βήματα πρόοδου. Αναφερθήκατε στις προτάσεις όσα ιδιαίτερα για τον BEPS. Πραγματικά εκεί περιλαμβάνονται πολλά ε, σωστά, όσο και απαραίτητα απολύτως. Αλλά σε ένα σημείο κάπως με έχετε απογοητεύσει γιατί δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιδράσει ή τι θέση έχει για τις προτάσεις του Κοινοβουλίου η Προεδρία. Εμείς ως πεμπτουσία του τάξε 1 ζητήσαμε δεσμευτικά νομοθετήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγίες, ακόμα και κανονισμούς ζητήσαμε που να ισχύουν και για τα 28 κράτη-μέλη με τρόπο δεσμευτικό, διότι έχουμε τον εξή φόβο ακριβώς η διαφορετική εφαρμογή των συστάσεων BEPS θα οδηγήσει σε ένα συνδυασμό 28 υπέρ ε, περίπλοκων φορολογικών συστημάτων που και πάλι θα έχουν παραθυράκια και δυνατότητες διαφυγής. Οπότε, σε μια εσωτερική αγορά ε, που γνωρίζει ελευθερία στην κυκλοφορία των κεφαλαίων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δεσμευτικά και ενία να εφαρμόζονται οι ε, κανόνες BEPS ε, με συνέπεια και με υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαγγείλει τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αλλά αν κατάλαβα καλά τον κύριο Μοσκοβισή, για την καινοτομία και τι ευρεσιτεχνίε τα έχει εξαιρέσει. Δηλαδή έχει πάρει τι αποστάσει τη, δεν θέλει να κάνει νομοθετικέ προτάσει, γιατί από ό,τι φαίνεται τα κράτη-μέλη δεν ε, δηλώνουν προθυμία ή δεν υπάρχει επαρκή προθυμία για να προχωρήσουμε σε μια κοινή νομοθεσία. Σε αυτό ακριβώ το σημείο χρειάζεται δουλειά να καλυφθούν τα κενά τουλάχιστον αυτό που αναλαμβάνω είναι η πέμπτουσία και της έκθεσης της Επιτροπής ΤΑΞ 1 που πέρασε με συντριπτικότατη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Με 508 ψήφους υπέρ, να δεν Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ Υπουργέ. Όλοι έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι αλλάζει η ε, ε, νοοτροπία ε, ο τρόπος με τον οποίο φορολογούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και όπως ισχύει και για τις τράπεζες, υπήρχε μια περίοδος προ Lehman Brothers και μετά Lehman Brothers. Όπως αντίστοιχα υπήρξε μια περίοδος όπου το τραπεζικό το θεωρεί το θεμητό, ενώ σήμερα θεωρείται αθέμητο, παντού όμως. Έτσι υπήρξε και μια περίοδος προ LuxLeaks και θα υπάρξει ένα μετά LuxLeaks και μάλιστα με έκπληξη είδαμε ότι όλες οι κυβερνήσεις μετά το LuxLeaks ε, άρχισαν να παίρνουν μέτρα. Εθνικά ή δεσμεύτηκαν να καταργήσουν κάποια καθεστώτα, να, να διαρθρώσουν την εφορία τους κτλ. Και μετά από την πίεση της κοινή νόμης και υπό την πίεση της κοινή νόμης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσα που ήδη είχε αρχίσει από το 2009 τις εργασίες έφεραν προτάσεις μια πρώτη οδηγία στην οποία αναφερθήκατε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα rulings πέρσι εγκρίθηκε και άλλες προτάσεις που έχουν έρθει τώρα. Εμείς χαρήκαμε για τη συνεργασία που αρχίσαμε πέρσι με τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και εξακολουθούμε να χαιρόμαστε και για τη συνεργασία που αρχίζουμε σήμερα μαζί σας. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Καταλάβατε φαντάζομαι ότι πέρα από τα αιτήματα και τις προτάσεις και τις υποδείξεις των συναδέλφων, εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη διαφάνεια. Επανέρχομαι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας και τη σχετική ομάδα, δύο είναι τα προβλήματα στην ουσία, στην πράξη. Ο τρόπος με τον οποίο διευθύνεται, αλλά και το επίπεδο στο οποίο συνεδριάζουν. Πριν από 20 χρόνια συστάθηκε στο δικό σας επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικό, υπουργών, και τις τρεις-τέσσερις πρώτες χρονιές λειτουργήσε σε πολιτικό επίπεδο, όπου και τα αποτελέσματα ήταν πολύ συγκεκριμένα όσο και πολύ θετικά και στη συνέχεια ε, συνεδρία σε διοικητικό επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων. Και αν λειτουργούσε σωστά, δεν θα καταλήγαμε ποτέ να έχουμε το LuxLeaks. Και τώρα το πρόβλημα θα πρέπει να το ξαναδούμε αλλιώ. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της διαφάνειας. Και αυτά που μας είπατε μας καθησύχασαν πάρα πολύ. Σας προτείνουμε λοιπόν, Υπουργέ, στο τέλος της Προεδρίας των κάτω χωρών να το ξαναπούμε. Για να κάνουμε ένα απολογισμό, να δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Voilà, Εάν euh, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα ε, κηρύξω τη λήξη της συνεδρίας της επόμενη. Να σας πω πότε είναι. Στις 14 Μαρτίου στις 3.30 λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Λήξη συνεδρίαση.